Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε. Ξεκινάει η σημερινή συνεδρίαση. Πρώτο σημείο συνήθω έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θεωρώ ότι είναι εγκεκριμένη. Περνάμε στο σημείο 2. Μία ανακοίνωση έχω σε ό,τι αφορά την έγκριση δύο προφορικών ερωτήσεων από του συντονιστέ τη Επιτροπή ΕΚΟΝ. Οι συντονιστέ τη 12 Νοεμβρίου ενέκριναν μια προφορική ερώτηση προ την Επιτροπή για την δίκαιη φορολόγηση στην ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία, BEPS 2. Η προφορική ερώτηση έχει διανεμηθεί στα μέλη στι 13 Νοεμβρίου. Επίση, ενέκριναν μια προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, πρόληψη της, ε, ε, των συγκρούσεων συμφερόντων κατόπιν ε, πρόσληψη. Η προφορική ερώτηση διανεμήθηκε στα μέλη στι 27 Νοεμβρίου. Και για τι ε, διαθεσμικέ διαπραγματεύσει, μια σύντομη ενημέρωση. Πρώτα απ' όλα για τα θέματα crowdfunding Στις 25 Νοεμβρίου είχαμε τον τρίτο γύρο τριμερούς διαλόγου ε, για τον βαθμό εναρμόνισης και το όριο των ε, μεμονωμένων προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από τις πλατφόρμες καθώς και το πεδίο του κανονισμού. Έχει επιτελεστεί πρόοδος στα βασικά θέματα αλλά υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να συζητηθούν ε, όλος ιδιαίτερο το θέμα της προστασίας των επενδυτών που θα συζητηθεί στην τέταρτο γύρο τριμερούς διαλόγου στις 11 Δεκεμβρίου. Ο δεύτερος τριμερής διάλογος είναι για την ταξονομία ο οποίος έλαβε χώρα στις 20 Νοεμβρίου. Την πλευρέ ε, στη διαπραγμάτευση ε, είχαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση, την πλατφόρμα για βιώσιμη χρηματοδότηση, ε, την ομάδα εμπειρογνωμόνων, τη κατεξοδότηση και εφαρμοστικέ πράξει και την εποπτεία. Εντελεχεί συζητήσει θα γίνουν για τι διαδικασίε μετάβαση και τη σχέση μεταξύ της ε, Δημοσιοποίηση και τη ταξονομίας. Μετά στι 27 Νοεμβρίου υπήρξαν περαιτέρω ανταλλαγέ απόψεων για τα τεχνικά κριτήρια ε, ελέγχου, τι οικονομικέ δραστηριότητε με σημαντικό αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τη ρήτρα αναθεώρηση. Έγινε μεγάλη πρόοδο στα άρθρα 1-4 μεταξύ των οποίων το πεδίο του κανονισμού και του ορισμού και στα άρθρα 5-12 συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών στόχων. Ο επόμενο γύρο τριμερού διαλόγου θα λάβει χώρα αύριο στι 3 Δεκεμβρίου. Και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις πάμε απευθείας στο βασικό θέμα για σήμερα. Νομισματικός διάλογος σε συνομιλία με την κυρία Λαγκάρτ. Καλωσορίζω την ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστή Λαγκάρτ στο ε, Κοινοβούλιο για τον τελευταίο γύρο του νομισματικού διαλόγου για φέτος, που όμως για την κυρία Λαγκάρτ είναι ο πρώτος. Θα θυμάστε ότι στις 23 Σεπτεμβρίου είχαμε την τελευταία ενημέρωση. Από την τελευταία φορά δεν έχει αλλάξει νομισματική ε, στάση ε, της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μέσα των πολιτικών μέτρων που εγκρίθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο συνεχίζουν να εγκρίνονται μέτρα για να συνεχιστεί ο ρυθμός ανάπτυξης που όμως χαρακτηρίζεται από βραδύτητα στην, ε, στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και την αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό οι κακές, συνθήκε κακές συνθήκες δανειοδότησης προς τα νοικοκυριά πρέπει να ε, μελετηθούν και θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιωθούν η ε, αντίσταση στις εγχώριες πιέσεις στις τιμές και η αντίσταση και μάλλον η μισοπρόθεσμη στόχη για τον πληθωρισμό της ΕΚΤ. Σήμερα η κυρία θα μας παρουσιάσει τη δική της προοπτική για τις μακροοικονομικές ε, προτεραιότητες καθώς και τις δύο προτεραιότητες των συντονιστών της Επιτροπής ΕΚΟΝ ε, όταν προετοίμαζαν αυτό το γύρο ε, νομισματικού διαλόγου, δηλαδή την αναθεώρηση τη νομισματική πολιτική και τη στρατηγική τη ΕΚΤ και το μέλλον για το χρήμα. Ε, κάναμε κάποια προπαρασκευαστική δουλειά για αυτό το θέμα με την ε, συνεισφορά πολλών μελών και τα έγγραφα είναι διαθέσιμα ε, στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση τη νομισματική πολιτική, μάλλον τη στρατηγικής πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζα, εκτιμούμε ότι από την τελευταία φορά το Σεπτέμβριο θα πρέπει να υπάρξουν κάποια βήματα προόδου που υπάρχουν διαφορετικέ απόψει για το επιθυμητό πεδίο και το μορφ, τη μορφή τη αναθεώρηση. Εγώ πιστεύω και έτσι ερμηνεύω ότι έχει και η άποψη που ε, επικρατεί εδώ, ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο ρόλο στο Ευρωκοινοβούλιο και σε αυτή την Επιτροπή όλο ιδιαίτερο στην όλη διαδικασία αναθεώρηση. Ελπίζω λοιπόν ότι η Πρόεδρο θα λάβει υπόψη το αίτημα αυτό. Ε, και έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε μαζί σα, πολλέ προσδοκίε από αυτή την πρώτη μα συζήτηση. Οπότε, κυρία Λαγκάρντα, σας δίνω το λόγο. Uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη. Τώρα ακούγεται. Oh. Αγωνιζόμαστε λοιπόν και προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι ακριβώς κάνουμε και ποια ακριβώς είναι η αποστολή μας και πώς τη φέρουμε σε πέρας. Όπως έλεγα και νωρίτερα, για μένα τις τελευταίες μέρες η πιο δυνατή στιγμή ήταν εκείνη όταν υπέγραψα ε, το πρώτο μου σημείωμα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και να ξέρετε ότι έχοντας ακούσει και από τον κύριο Τρισέ πόσο σημαντική εκείνη η στιγμή, και όταν ακούω από φίλους και συγκινείς που μου λένε ότι θέλουν, γιατί αυτό ακριβώ έκανα βασικά το πρώτο χαρτονόμισμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι περισσότερο μου λένε ότι το θέλουν να γίνει πραγματικότητα και να το δούνε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μην ξεχνάμε ότι και εμείς είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το ευρώ. Στην ε, περιοχή του ευρώ λοιπόν, στην ευρωζώνη, η αξιοπιστία του κοινού νομίσματος αυξήθηκε. Βρισκόμαστε σε ένα χαμηλό του 62% το 2013, κατά τη διάρκεια της κρίσης δηλαδή, και έχουμε φτάσει στο υψηλότερο ποτέ ποσοστό που είναι 76% σήμερα. Η εμπιστοσύνη λοιπόν στους θεματοφύλακες του ευρώ, που είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επίσης αυξήθηκε, όχι βέβαια τόσο πολύ όσο αυξήθηκε και για το ευρώ. Οι προκάτοχοί μου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν πάρα πολύ προσεκτική για αυτά και έκαναν τα πάντα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Οι πρακτικές λογοδοσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξελίχθηκαν, όπως επίσης και η στρατηγική της επικοινωνίας και η διαφάνεια της ΕΚΤΑ ε, τα ηθικά, ηθική, η χρηστή διακυβέρνηση, όλα αυτά τα πλαίσια εναρμονίστηκαν, ενισχύθηκαν και επεκτάθηκαν σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι η σχέση με τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους των οποίων την υπηρεσία βρισκόμαστε. Και προσπαθούμε να βελτιώσουμε κυρίως τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε με το γενικό κοινό. Και γι' αυτό ακριβώς ο δικός σας ο ρόλος που είσαστε ευρωβουλευτές που είσαστε μέλη αυτής της Επιτροπής είναι τόσο πολύ σημαντικός. Γιατί εσείς φροντίζετε να ακούγεται η φωνή των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά επίσης να ακουστεί και η φωνή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στον κόσμο. Η επικοινωνία για μένα είναι προ δύο κατευθύνσει και είναι πολύ σημαντική για τη δημοκρατία που αποτελεί και βασική αρχή τη Ευρώπη, Και σε αυτό το πνεύμα λοιπόν είναι που θα προσεγγίσω και εγώ την ακρόαση αυτή και όλε τι επόμενε που προβλέπω να έχω μαζί σα τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ε, πρώτα απ' όλα από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη, στην οποία αναφερθήκατε και εσείς στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις και μετά θα έρθω στις δύο ερωτήσεις για τις οποίες μου ζητήσατε σχόλια. Η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη παραμένει αδύναμη. Το ΕΠ αυξήθηκε μόνο 0,2% από το ένα τρίμηνο στο επόμενο, το τρίτο τρίμηνο δηλαδή το 2019. Και αυτή η αδυναμία κυρίως βασίζεται σε παγκόσμιους παράγοντες. Η παγκόσμια οικονομία παραμένει επίσης αδύναμη και αβέβαιη και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται η ζήτηση στην Ευρωζώνη για αγαθά και υπηρεσίες, αλλά επηρεάζει επίσης και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Και καθώς είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτές τις παγκόσμιες εξελίξεις και ο κατασκευαστικός τομέας έχει επηρεαστεί κατά πολύ και επηρεάζονται βέβαια και άλλα τμήματα της οικονομίας με τελευταίες εκθέσεις να λένε ότι και οι υπηρεσίες επηρεάζονται. Παρ' όλα αυτά όμως, η κατανάλωση έχει προχωρήσει καλά, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας επίσης βελτιώνονται και ενθαρρύνονται οι καταναλωτές να δείχνουν εμπιστοσύνη και να δαπανούν. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για την οικονομία μας. Τώρα, οι ε, δυναμία στην οικονομική δραστηριότητα έχει επηρεάσει όμως τις εξελίξεις των τιμών. Και ξέρετε ότι αυτή, αυτή η υποτονικότητα είναι για μας κάτι πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ο πληθωρισμός ήταν 1% τον Νοέμβριο. Και αν ε, κοιτάξουμε έρευνες που βασίζονται στην αγορά ή τις προπτικές του πληθωρισμού, ε, βρισκόμαστε σε ιστορικά πάρα πολύ χαμηλά. Οπότε, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα σε ένα δύναμο οικονομικά περιβάλλον για να σεβαστεί το ρόλο τη που είναι η διατήρηση σταθερότητα των τιμών. Πρώτα απ' όλα, η νομισματική πολιτική μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά ακόμα και αν η ανάπτυξη είναι χαμηλή εξαιτία εξωτερικών παραγόντων και μπορεί να το κάνει αυτό διασφαλίζοντα ευνοϊκέ συνθήκε χρηματοδότησης για όλου του τομεί τη οικονομία και προσφέροντα επίση προβολή ε, των συνθηκών ε, αυτών και να φροντίσει να τις διατηρεί και στο μέλλον. Έτσι λοιπόν έχουμε πιστώσει σε όρους κάπως ικανοποιητικού. Συνεπώς, τα νοικοκυριακή επιχειρήσεις μπορούν να καταναλώσουν και μπορούν να επενδύσουν περισσότερο. Αυτή η στήριξη για την εσωτερική ζήτηση ενισχύει επίσης κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος βεβαίω και είναι εκείνος που απασχολεί περισσότερο εργατικό δυναμικό στην οικονομία μας. Και αυτό με τη σειρά του βοηθάει να προστατευτούν οι θέσεις απασχόλησης, τα εισοδήματα και να διατηρηθεί η κατανάλωση με αντιστάθμιση δηλαδή των εξωτερικών αρνητικών παραγόντων. Αυτός ο μηχανισμός σήμερα λαμβάνει χώρα. Υπάρχει αντοχή των υπηρεσιών μέχρι τώρα και αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η απασχόληση έχει επηρεαστεί πολύ λίγο από την επιβράδυνση στον τομέα της μετοποίησης. Και εξαιτία αυτών των αδύναμων προοπτικών, το Δικητικό Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έλαβε κάποιε αποφάσει τον ε, Σεπτέμβριο που μα πέρασε, προκειμένου να φροντίσει οι συνθήκε χρηματοδότηση να παραμείνουν ευνοϊκέ. Όπω θα θυμόσαστε, γιατί ο προκάτοχός μου, ο κύριο Στράκης, σα τα είπε στι 23 Σεπτεμβρίου, το Δικητικό ε, Συμβούλιο αποφάσισε τότε ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει μείωση του επιτοκίου διευκόλυνσης καταθέσεων. Μειώθηκε δηλαδή αυτό στο μείον 0,5%. Το δεύτερο κομμάτι στο πακέτο είναι να αρχίσει πάλι η αγορά στοιχείων ενεργητικού. Το τρίτο ήταν να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο και τα επιτόκια αλλά και την αγορά, το πρόγραμμα δηλαδή αυτό. Το τέταρτο είναι να φροντίσουμε για τις στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότησης, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο χρηματοδοτεί την οικονομία μας, το TLTRO, να γίνει ακόμα πιο ελκυστικό το πρόγραμμα αυτό και το τελευταίο ήταν να φροντίσουμε να εισάγουμε ένα ε, νέο σύστημα ε, ανταμοιβή ε, των τραπεζών που διακατέχουν μεγαλύτερα κεφάλαια. Τα μέτρα αυτά λοιπόν θα λειτουργήσουν χέρι-χέρι, προκειμένου τα επιτόκια να διατηρηθούν για όλες τις λεκτικότητες γύρω από ένα επίπεδο που να συνάδει με την διευκολυντική μας πολιτική. Τώρα, τα αρνητικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Τράπεζας επηρεάζουν με τη σειρά τους τα επιτόκια, τα βραχυπρόθεσμα και τα μέσο πρόθεσμα, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα να βοηθήσουν τις τράπεζες να δανείζουν. Εκ με αυτό, η καθαρά αγορά ομολόγων βοηθάει επίσης τις αποδόσεις τις μεσοπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες, κάτι το οποίο βοηθάει μακροπρόθεσμα δάνεια, τα οποία συνήθως γίνονται από τις τράπεζες στα νοικοκυριά. Οι πιο ελκυστικές λοιπόν συνθήκες του περίφημου TLTRO βοηθούν οι πιστώσεις των τραπεζών να κυκλοφορούν και να φτάνουν υπό ευνοϊκές συνθήκες στους καταναλωτές. Και επικεντρωθήκαμε επίσης σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στα νοικοκυριά. Συγχρόνως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε το Σεπτέμβριο δείχνοντας ότι είναι έτοιμο να παρακολουθήσει και όλες τις παρενέργειες της νομισματικής πολιτικής. Αυτό το νέο σύστημα λοιπόν δύο βαθμίδων ε, για την ε, ανταμοιβή ε, των τραπεζών που διακατέχουν μεγαλύτερα κεφάλαια, βοηθάει την ρευστότητα στο ευρωσύστημα παρά τα αρνητικά επιτόκια στις καταθέσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να έχουμε διευκολυντική πολιτική και στη συνέχεια για την οικονομία μας. Αυτή λοιπόν η πολιτική της έκτη διευκολυντική είναι εκείνη η οποία βοήθησε την ανάκαμψη και την συνεχίζουμε. Και όπως αναφέρεται στις κατευθύνσεις γραμμές της ΕΚΤ, η νομισματική πολιτική θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία και να ανταποκρίνεται σε μελλοντικού κινδύνους, ευθυγραζόμενη με τον, το κύριο καθήκον της που είναι η σταθερότητα των τιμών. Και θα συνεχίσουμε βεβαίως να παρακολουθούμε τις παρενέργειες των πολιτικών μας. Όπω σα επιβεβαίωσα και την προηγούμενη φορά όταν ήμουν εδώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένει αποφασισμένη να τηρήσει τις υποχρεώσεις της και την εντολή της, να συμμορφωθεί προς την εντολή της. Κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό για τη σταθερότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης και για την ευημερία των πολιτών στην Ευρωζώνη. Αλλά μου ζητήσατε επίση να συζητήσω μαζί σα και δύο στοιχεία κλειδί που κατά τη γνώμη μου είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα και που αντιμετωπίζει η νομισματική μας πολιτική. Και μου ζητήσατε κυρίως να μιλήσω για την στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Η αναθεώρηση της στρατηγικής μας αυτής θα ξεκινήσει σύντομα. Όπως θα γνωρίζετε, μια στρατηγική νομισματικής πολιτικής δεν είναι κάτι πρωτάκουστο είναι κάτι το οποίο γίνεται από πολλές κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο με διαφορετικούς ρυθμούς, διαφορετικές στιγμές, διαφορετικό βηματισμό. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η Fed ε, κάνει μια τέτοια αναθεώρηση και θα την ε, ολοκληρώσει, αυτήν η οποία ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο περίπου, θα την ολοκληρώσει στο δεύτερο εξάμενο του 2020. Έπειτα, Κεντρική Τράπεζα του Καναδά. Επίσης, έχει τέτοιες αναθεωρήσεις στρατηγικής κάθε πέντε χρόνια, έτσι ώστε να είναι σίγουρη ότι συμμορφώνεται προς την εντολή της. Στη δικιά μας την περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λοιπόν, είχε μια τέτοια αναθεώρηση το 2003, πριν από 16 ολόκληρα χρόνια δηλαδή. Και αυτά τα 16 χρόνια πολλά έχουν συμβεί. Το μακροοικονομικό τοπίο βέβαια έχει επηρεαστεί από την μεγάλη οικονομική κρίση του 2008 και τις κρίσεις δημοσίου χρέους που ακολούθησαν. Πιο πρόσφατα, το τοπίο αυτό επηρεάζεται επίσης από το χαμηλό πληθωρισμό παντού στον κόσμο, λίγο πολύ σίγουρα στις πιο αναπτυγμένες οικονομίες. Συγχρόνω όμω, υπάρχουν και νέε προκλήσεις μπροστά μας, δημογραφικές αλλαγές, η γύρανση του πληθυσμού, κυρίως στι αναπτυγμένες οικονομίες, αλλά επίση και τεχνολογικές αλλαγές ιδίω ε, όταν αυτές είναι πιο γενικές και έχουμε βέβαια και την κλιματική αλλαγή η οποία κυριαρχεί τις συζητήσεις σήμερα και απασχολεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον και έχουν κάποιες πολιτικές ευθύνες. Έπειτα η συμβατική σοφία που εφαρμόζαμε μέχρι τώρα επίσης έχει βρεθεί στα όρια της και η πολιτική μας χρειάστηκε να βρεθεί σε χαρτογράφητα νερά. Όλα αυτά λοιπόν ζητούν από εμά να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μας και να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε καλύτερα να τα βγάλουμε πέρα. Και πράγματι ένα ερώτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τις κεντρικές τράπεζες και το συζητούν και άλλοι αλλά και εμείς φυσικά στην ΕΚΤ είναι πώς να καθορίσουμε καλύτερα τους μεσοπρόθεσμους στόχους της νομισματικής πολιτικής έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προοπτικές και οι ε, προβλέψεις όντως ε, θα υλοποιηθούν. Σε μια κατάσταση σαν τη σημερινή Πάντως, όπου η οικονομία έρχεται αντιμέτωπη με πολλές δυσκολίες και εμπόδια, δεν μπορεί αυτό να επιτευχθεί τόσο καλά όσο πριν από την κρίση. Και όλοι προσπαθούμε να δούμε πώς οι μακροπρόθεσμες τάσεις, τις οποίες αναφέρθηκα πριν, θα επηρεάσουν τελικά το δικό μας ενεργητικό και πώς θα ελέγξουμε την κατάσταση. Τώρα, θα ήταν βέβαια πρόωρο και θέτε και αντιπαραγωγικό κατά τη γνώμη μου τώρα να σας ε, πω ε, πώς ακριβώς θα έχει αυτή η αναθεώρηση της ε, στρατηγικής μας. Στο κάτω-κάτω ακριβώς αυτό προσπαθούμε να δούμε. Να καταλήξουμε σε κάτι ολόκληρο το Συμβούλιο και να ανοίξουμε νέες οδούς για διάλογο με όσους ενδιαφέρονται για το θέμα. Αυτό σημαίνει εμπειρογνώμονες, και εσείς ε, είπατε ότι και εσείς συζητάτε με πυρογνώμονες. Σημαίνει επίσης ότι στη συζήτηση αυτή θα συμμετάσχετε και εσείς διότι εσείς θα μεταφέρετε σε μας τις απόψεις που ακούτε από τους πολίτες σας. Και αυτή είναι μια επικοινωνία στην οποία πιστεύω πραγματικά και νομίζω ότι θα έχει θέση σε αυτή τη στρατηγική. Τώρα με ποιο ρυθμό, πού, πώς, ε, πότε, ε, με ποιο ρυθμό κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο για το οποίο θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας. Αλλά δεν πρόκειται εδώ να αποφασίσω για κάτι τέτοιο, γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εκείνο το οποίο θα αποφασίσει για το πώς ακριβώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία και ποιο θα είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα έχουμε την αναθεώρηση της στρατηγικής μας. Έπειτα, εκπρόσωποι της κοινωνίας επίσης θα πρέπει να έχουν λόγο και θα ήθελα να τους ακούσω για την νομισματική μας πολιτική και για το πώς θα συμμορφωθούμε προς την εντολή μας. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι θα εφαρμόσουμε δύο αρχές. Η πρώτη είναι σε βάθος ανάλυση και η δεύτερη είναι να είμαστε ανοιχτοί. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε χρόνο για προβληματισμό και για να ακούσουμε όλους τους εταίρους στους οποίους αναφέρθηκα πριν. Τώρα, οι προκάτοχοί μου μου ανέφεραν ότι προηγουμένως το 2003 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας ε, πρότεινε ένα φόρουμ για διάλογο που εμπλουτίστηκε από τις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη προετοιμαστεί. Η ΕΚΤΕ σίγουρα υποφελήθηκε από τις συζητήσεις αυτές πριν από 16 χρόνια, τότε που είχε την προηγούμενη της αναθεώρηση για την νομισματική της στρατηγική. Αυτή τη φορά δεδομένου ότι η επικοινωνία είναι πιο ζωντανή, ε, δεδομένου ότι έχουμε νέα μέσα επικοινωνίας, σίγουρα μπορούμε να ανοίξουμε το πεδίο ακόμα περισσότερο και ότι θα έχουμε ακόμα πιο ζωντανές ανταλλαγές απόψεων και πλούσιο διάλογο μεταξύ μας. Αλλά βλέπω να είναι δικιά μου ευθύνη, μια που είμαι πρόεδρος της ΕΚΤ, να έρχομαι να αναφέρω σε εσά και να ζητάω τη γνώμη σας. Όπως είπα, άπαξ και το Διοικητικό Συμβούλιο της εκτε. έχει εντοπίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μας, θα ξανέρθω για να πούμε περισσότερα. Τώρα, το δεύτερο θέμα που μου ζητήσατε να συζητήσουμε σήμερα είναι το μέλλον του χρήματος, όπως το λέμε. Πράγματι, οι κεντρικές τράπεζε βρίσκονται σε έναν χώρο που συνεχώς αλλάζει. Οπότε δεν θα έπρεπε απλώς να προσπαθούμε να προλάβουμε τις μελλοντικέ τάσεις, αλλά και να τις διαμορφώσουμε, για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε μια καλή ανάλυση του κόστους και του ωφέλους. Το περιβάλλον επίσης των οικονομικών υπηρεσιών επίσης τροποποιείται και επαναστατικά πολλές φορές. Υπάρχει ζήτηση από τον κόσμο. Γίνονται συζητήσεις για τα λεγόμενα σταθερά νομίσματα που οδηγούν σε αλλαγές και πολύ περισσότερο στο μέλλον. Αυτό το, ε, αυτές οι εξελίξεις βέβαια μπορεί να αλλάξουν ε, το τοπίο για τα νομίσματα και να οδηγήσουν ακόμα και σε αστάθεια και να επηρεάσουν πολλά πράγματα. Αλλά να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Πέρυσι και μάλιστα το θυμάμαι όταν ήμουν μαζί σας στην ακρόασή μου εδώ, θυμάμαι ότι ανέφερα κάτι. Βέβαια, σας ανέφερα το tips και σίγουρα το ξέρατε κι εσείς, εγώ το έμαθα το tips, ξέρω τώρα περισσότερα από όσα ήξερα τότε. Το tips λοιπόν είναι ένας διακανονισμός άμεσων πληρωμών. Ήταν κάτι που δεν γνωρίζαμε τότε αρκετά, γιατί συνέβαινε ε, στα παρασκήνια μεταξύ των τραπεζών έτσι ώστε να γίνονται απευθεία πληρωμές μεταξύ των τραπεζών 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο. Συμβαίνει στα, στα παρασκήνια αλλά επιτρέπει ε, άμεσες πληρωμές μεταξύ τους και είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται ε, σε αυτό που το κοινό ζητάει, άμεσες πληρωμές ώστε όσοι έχουν κάποιο λογαριασμό στην Ευρώπη να μπορούν να κάνουν αυτές τις συναλλαγές απευθείας. Προσφέροντας ε, λοιπόν στο χρήμα της Κεντρικής Τράπεζας τις συναλλαγές αυτές, αυτό βοηθάει τις συναλλαγές του κόσμου σε καθημερινή βάση. Δεν είναι κάτι βέβαια που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στις τράπεζες ακόμα, γιατί έχουν και τα δικά τους συστήματα, αλλά ελπίζουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί όλο και περισσότερο και θα διαδοθεί επαρκώς για να διευκολυνθούν οι συναλλαγές και να είναι περισσότερο ασφαλείς. Δεύτερον, από το 2016 η ΕΚΤ επίση εξετάζει και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, κυρίως τις λεγόμενες Distributed Ledged Technologies για τις ε, υποδομές μαζί με την Τράπεζα της Ιαπωνίας έχουμε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Στέλλα και το οποίο βοηθάει να υπάρχουν πιο φτηνές και πιο γρήγορες και περισσότερο ασφαλείς συναλλαγές. Αλλά σημαίνει επίσης ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε και τους κινδύνους που έρχονται μαζί. Η καινοτομία και τα stable coins είναι κάτι από το οποίο μπορούμε να υποφεληθούμε επόσον οι κίνδυνοι είναι ελάχιστοι. Και αυτό θα το πετύχουμε με ρυθμίσεις. Και εδώ είναι που έρχεστε εσείς. Συνεπώς πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε το χρυσό κανόνα της εποπτείας. Δηλαδή, ίδιο ίδιοι, ίδιο κλάδοι, οι ίδιοι κίνδυνοι, οι ίδιοι κανόνες, όποια και είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείτε. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα stable coins δεν μειώνουν την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα των πληρεμών ή τη σταθερότητα του νομισματικού συστήματος. Και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό για coins, τα οποία χρησιμοποιούνται διεθνώς. Η ομάδα εργασίας G7 υπό τον Benoit Κερέ έχει προβεί σε συγκεκριμένες συστάσεις για την ανάπτυξη μιας συνολικής και παγκόσμιας προσέγγισης ρυθμίσεων. Όπως έγινε και με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, το περίφημο GDPR, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι μπορεί να δείξει το δρόμο. Στην ίδια γραμμή, με διεθνείς προδιαγραφές και συστάσεις και εμείς, και εσείς βέβαια είσαστε συνομοθέτες, μην το ξεχνάμε, πρέπει να αναπτύξουμε ε, μία ρύθμιση με σωστή ισορροπία. Από τη μια μεριά να έχουμε την καινοτομία και από την άλλη μεριά τους κινδύνους. Να στηρίξουμε βέβαια την καινοτομία, αλλά να προστατεύσουμε από κινδύνους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν είναι έτοιμη να παίξει το δικό της ρόλο και συνεργάζεται και με άλλες κεντρικές τράπεζες και τις εθνικές αρχές προς το σκοπό αυτό. Επίσης αναθεωρούμε και το πλαίσιό μας όσον αφορά ε, καινοτόμες μεθόδους για πληρωμές και έτσι παρακολουθούμε μία προσέγγιση βάσει αναλογικότητας ε, και βασισμένου στους κινδύνους. Εμείς θα λειτουργήσουμε ως καταλήτες και θα βοηθήσουμε όλες τις πλευρές ώστε να καταλήξουμε σε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών. Επίσης, παίζουμε το ρόλο μας με πλήρη ανεξαρτησία αξιολογώντας τα ψηφιακά ε, νομίσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες και γενικότερα για την οικονομία. Ένα ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας θα μπορούσε να επιτρέπει στους πολίτες να το χρησιμοποιούν απευθεία καθημερινά. Αλλά ανάλογα με το πώς θα σχεδιαστεί, ένα τέτοιο ψηφιακό νόμισμα μπορεί να ελοχεύει και κινδύνου. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο προχωράει νομισματική πολιτική και μετακυλείται στην πραγματική οικονομία. Επίσης θα μπορούσε να έχει και επιπτώσεις στη λειτουργία του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και τη σταθερότητά του. Οπότε ε, το ζήτημα του νομίσματος κεντρικής τράπεζας, του ψηφιακού δηλαδή, χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Πάντως θέλουμε να καταλήξουμε σε πληρωμές ολοκληρωμένες με καινοτομία και ασφαλής. Αυτό θα είναι προ όφελο όλων και θα ενισχύσει διεθνώ ακόμα περισσότερο και το ευρώ. Συνεπώ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ μέλη τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Οι εκλογέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδειξαν σαφέστατα ότι ο κόσμος περιμένει φιλόδοξες απαντήσεις από τη δικιά σας την πλευρά. Πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες αυτές συνεργαζόμενοι, γιατί μόνο έτσι θα ανακτηθεί η του κόσμου στην Ευρώπη, στο ευρώ και στην ΕΚΤ. Ο Ζάμονε είπε κάποτε ότι όλοι είμαστε φιλόδοξοι. Το θέμα είναι αν κάποιος είναι φιλόδοξος για να είναι φιλόδοξος ή αν είναι φιλόδοξος για να κάνει πράγματα. Λοιπόν, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στην ΕΚΤ εμείς είμαστε φιλόδοξοι για να κάνουμε πράγματα και να τα κάνουμε από κοινού με άλλου κάθε φορά που αυτό καθίσταται εφικτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σα ευχαριστώ κυρία Λαγκάρτ. Περνάμε στι ερωτήσει ε, για ανταλλαγή απόψεων. Σα παρακαλώ να θυμάστε ότι έχετε συνολικά πέντε λεπτά για την ερώτηση και την απάντηση. Δύο ερωτη... λεπτά για την ερώτηση, τρία λεπτά για την απάντηση. Ε, Λίδια Περέιρα από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Κυρία Λαγκάρτ, καλώς ήρθατε στο Κοινοβούλιο ξανά και για πρώτη φορά ως Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σας καλωσορίζω στο Κοινοβούλιο, στα πρωτογαλλικά. Οι πολίτες θέλουν μια οικονομία ακριβίας, με ένα ευρώ ισχυρότερο, το οποίο να εξυπηρετεί την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Η νομισματική πολιτική είναι καθοριστικής σημασίας και η πολιτική χαμηλών επιτοκίων είναι πρόσδεκτα μέτρα. Όμως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τους τρέχοντες λογαριασμούς σε ρευστότητα πάνω από 20 δις με χώρες που έχουν σοβαρό δημόσιο χρέος και είναι σε ευπαθή κατάσταση. Πρέπει να αναζητήσουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Σε άλλες όμως χώρες είναι πολύ κοντά στο να βρεθούν κοντά στα όρια των στοιχείων ενεργητικού που έχουν οριστεί. Κυρία Λαγκάρντ, πέρσι είδαμε ότι οι δημόσιες επενδύσεις στην Ευρωζώνη είναι κάτω των επιπέδων, είναι χαμηλότερο των επιπέδων πρώτης κρίσης. Γι' αυτό θα πρέπει τα δημοσιονομικά των κρατών να φτάσουν σε τέτοια επίπεδα που να επιτρέπουν επενδύσεις. Σε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Κύπρος, οι δημόσιες επενδύσεις είναι, είναι κοντά στο 2%. Και Υπάρχουν ε, σοβαρές κρατικές επενδύσεις που ε, πρέπει να γίνουν για να ανταποκριθούμε στις επενδύσεις των πολιτών. Υπάρχουν ένα ελάχιστο επίπεδο επενδύσεων, οπότε τι ρόλο μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τι μπορεί να γίνει για την κατάσταση των πολιτών σε σχέση με το χρέος και την ε, γενικότερη πολιτική για την ενίσχυση των κρατικών επενδύσεων. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, που κατά τη γνώμη μου έχει ως αντικείμενο ένα πολύ σημαντικό θέμα, τις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα. Για μένα και πολλούς από όσους το διάβασαν ήταν συναρπαστικό να διαπιστώσουμε το συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την ε, έλλειψη επενδύσεων. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει μια κεντρική τράπεζα. Καταρχάς πρέπει να αναρωτηθεί. Ποια είναι η εντολή μου. Η εντολή της είναι σταθερότητα των τιμών που καθορίστηκε το 2003 υπό την στρατηγική αναθεώρηση που έγινε τότε ως κοντά αλλά κάτω από το 2%. Μια κεντρική τράπεζα λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της και αυτά που μπορεί να έχει στη διάθεσή της για να πετύχει τον στόχο αυτό. Την σταθερότητα των τιμών δηλαδή που περιγράφεται στην εντολή της. Η διευκόλυνση επενδύσεων, η πρόσβαση νοικοκυριών και επιχειρήσεων ε, σε κεφάλαια για να μπορέσουν να επενδύσουν είναι μία από τις βασικές ε, ανταποκρίσεις που μπορεί να προσφέρει μια κεντρική τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την κρίση και μετά πάντα προσπαθούσε να παρέχει τα εργαλεία αυτά ώστε να διευκολύνει και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις. Αυτό το κάνει με βάση τα δεδομένα, τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της και θα πρέπει να συνεχίσει να το κάνει αυτό εφόσον οι πληροφορίες δείχνουν συνεχή επιβράδυνση της οικονομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Φερνάντες από το S&D. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, Πρόεδρε. Έχω μία απλή ερώτηση. Στις σημερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ε, σε ποια ημερομηνία τηρείτε την εντολή σας. Δεν είμαι βέβαιη ότι κατάλαβα την ε, ερώτηση. Θέλετε προβλέψεις όσον αφορά τον πληθωρισμό για τη δικιά σας ε, ευθύνη δεν είναι αυτή. Νομίζω ότι κανείς δεν θα τολμούσε να κάνει προβλέψεις με συγκεκριμένο νούμερο όταν θα λήξει το εντολή όπως με ρωτήσατε, δηλαδή σε 8 χρόνια από τώρα ποιος θα είναι ο πληθωρισμός ή ποιο θα είναι, ποια θα είναι επιτόκια ανάπτυξη. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό και προσπαθούμε να βρούμε νέα μέσα και θα τα εξετάσουμε και σίγουρα όχι μόνοι μου βέβαια, εννοείται και ούτε μόνο ένα μέσο, αλλά στόχος μας είναι ακριβώς να καθορίσουμε με την αναθεώρηση τη νέα μας στρατηγική. Όλα τα μέλη της ΕΚΤ και το προσωπικό, οι εμπειρογνώμονες δηλαδή, εξετάζουν την εντολή μας που τώρα λέει κοντά αλλά κάτω από το 2%. Σε αυτό εμένουμε τώρα. Και αυτό προσπαθούμε όλοι να κάνουμε. Αλλά τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά όταν θα έχει γίνει η αναθεώρηση. Ωραία, δεν έχετε εσείς καμία ημερομηνία για πρόβλεψη. Στις προπτικές θα έχετε φαντάζομαι την ημερομηνία πότε πιστεύετε ότι θα είσαστε στο 2%. Απάντηση. Όσο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Και έχω και άλλη ερώτηση, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ε, συνεχίζω ισπανικά. Καταλαβαίνω λίγα ισπανικά, λέει η κυρία Λαγκάρτ. Ωραία. Λοιπόν, αναφερθήκατε στην αναθεώρηση του στρατηγικού πλαισίου της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Είναι κάτι για το οποίο σας ρώτησα και στην ακρόαση που είχαμε μαζί σας, εν ώψη του ορισμού σας. Και είχατε πει τότε ότι είναι νωρί για να πούμε προς τα πού θα πήγαινε αυτή η αναθεώρηση της στρατηγικής, της νομισματικής πολιτικής. Θέλω όμως να σας ρωτήσω για την τωρινή νομισματική πολιτική. Πότε πιστεύετε ότι ο σημερινός στόχος του 2 ή κάτω από 2% θα μπορέσει να θεωρηθεί συμμετρικός στόχος ή να μην θεωρηθεί συμμετρικός στόχος. Πότε νομίζετε ότι θα έχουμε μια απάντηση γι' αυτό. Η κυρία Λαγκάρ, το θέμα της συμμετρίας είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητηθεί στα πλαίσια της αναθεώρησης της στρατηγικής μας. Και η ΦΕΔ το κάνει το ίδιο στη δικιά της αναθεώρηση στρατηγικής και είναι κάτι που και ο προκάτοχός μου το είχε πει, ο πρόεδρος Ντράγκη, ότι υπάρχει μια συμμετρική φύση. Τώρα, δεδομένου ότι αναθεωρούμε ε, κάποια στοιχεία που σχετίζονται με το στόχο μας σταθερότητας τιμής, σίγουρα η έννοια της συμμετρίας θα αποτελέσει και αυτή μέρος της αναθεώρησής μας. Εξαρτάται τι στοιχεία κοιτάει κανείς. Αν ε, κοιτάει ένα εύρος, μια ευελιξία, έναν ώρα αναφορά κτλ. Πρέπει να αναρωτηθεί κανείς πάντα για την συμμετρία. Οπότε αυτή είναι μια άσκηση που θα λάβει χώρα. Δεν λέω για το τώρα, λέω ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη μελλοντική μας συζήτηση. Αυτό. Ευχαριστώ. Η Στεφανή Κουρτένα, από το Ρινιού. Κυρία Πρόεδρε, και πάλι ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Μεταξύ των πολυάριθμων δυσκολίων που θα έχει να αντιμετωπίσει η ΕΚΤ υπάρχουν δύο βασικέ προκλήσει. Η μία λίμωνο είναι πολύ ε, κλασική. Η ισότητα ανδρών και γυναικών, ιδίω το διορισμό των διευθυντών σε νομασματικού και οικονομικού φορεί και ε, θα θέλαμε να μην βλέπουμε πάντα αυτή τη φωτογραφία που είδαμε και πρόσφατα, όπου ήσασταν μόνοι, η μόνη γυναίκα στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Διευθυντών. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, θα, είσαστε, θα ήσασταν έτοιμοι να προβλέψουμε υποχρεωτικό κανόνα, βάσει του οποίου όλοι οι μελλοντικοί διορισμοί θα περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και μια γυναίκα ε, μαζί με έναν άντρα ταυτόχρονα, όπως πρότεινε πρόσφατα και η κυρία Ούρσουλα Φοντερ και μετά πρέπει να δούμε και τη δεύτερη πρόκληση, την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Την περασμένη εβδομάδα 164 ε, εμπειρογνώμονε και με κυβερνητικέ οργανώσει ζήτησαν από την ΕΚΤ να κάνουν ό,τι μπορεί για να επιταχυνθούν οι προσπάθειε καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών. Και αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα τη ε, επιθυμία τη κοινωνία των πολιτών να αναπτύξει σχέσει με την ΕΚΤ και να την λαμβάνουν και σοβαρότερα υπόψη για να καλλιεργηθεί ένας διάλογος, όπως το τονίσατε και πρόσφατα, αλλά και στην ακρόασή σας τον Σεπτέμβριο. Είναι σημαντικό και να αμοιβαία τα ωφέλη του να υπάρχει ένας ενεργός και ζωντανός διάλογος με την κοινωνία των πολιτών. Το είχατε πει και το Σεπτέμβριο, η πείρα σα θα είναι εδώ πολύτιμη. Είστε έτοιμοι να την ανανεώσετε αυτή την εμπειρία που ήδη έχετε με νέα παραδείγματα και να ε, συμπαρασύρεται την κοινωνία των πολιτών σε αυτή την κοινή προσπάθεια για να υπάρξει μια μετάβαση, μια καταπολέμηση, προσπάθεια καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση που έχει δύο πτυχές, δίπτυχη ερώτηση και θα προσπαθήσω να τις απαντήσω διαδοχικά. Πρώτη ερώτηση η καλύτερη εκπροσώπηση, σε εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών και κυρίως το να υπάρξουν περισσότερες γυναίκες στους οικονομικούς οργανισμούς. Ε, αυτόν τον αγώνα τον δίνω εδώ και πολλά χρόνια, θα συνεχίσω και πραγματικά με πολύ μεγάλη αισιοδοξία καλωσορίζω το δικό σας το ρόλο προσωπικά σε αυτή τη διαδικασία. Σήμερα το Συμβούλιο Διευθυντών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελείται ε, από 25 άτομα, εκ των οποίων 24 είναι κύριοι. Πολύ τους αγαπώ και πολύ τους συμπαθώ γενικώ τους άνδρες, Όμω η εκπροσώπηση αυτή προφανώ δεν είναι φυσιολογική και δεν αντικατοπτρίζει την κοινωνία μα. Και πραγματικά ελπίζω η κατάσταση αυτή να αλλάξει και να αλλάξει θετικά, ώστε να λαμβάνει υπόψη καλύτερα το σε τι είδου κοινωνία ζούμε. Δυστυχώ υπάρχουν κάποια στοιχεία που δεν ε, περνάνε από το δικό μου το χέρι, ούτε από την ΕΚΤ. Διότι όπω τα ξέρετε, από ε, του 25, οι 19 είναι διευθυντέ τη Κεντρική Τράπεζα του συστήματο που ονομάζουμε Ευρωσύστημα, το οποίο το λέω με μεγάλη συμπάθεια και αισθήματα φιλία απέναντί του. Είναι όλοι άνδρε, είναι όλοι κύριοι. Ε, δεν είναι στο χέρι μου, δεν είναι κάτι που είναι στην εξουσία μου, αλλά πιέστε τι εθνικέ αρχέ των χωρών από τι οποίε προέρχεστε για να γίνουν και γυναίκε αυτέ που είναι διευθυντρίε των κεντρικών τραπεζών. Εγώ ξέρω κάποιε υποψήφιε, θα μπορούσα, αν σα ενδιαφέρει, να σα δώσω τα ονόματα. Για του υποψηφίου. Το να έχουμε καταρχήν τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο από κάθε φίλο μου φαίνεται μια πολύ σωστή πρακτική. Θα το πω εγωιστικά και θα κάνω εδώ μια εξαίρεση, διότι ξέρω ότι αύριο θα περάσουν από ακρόαση δύο υποψήφοι. Ένας άντρας και μια γυναίκα και που είναι υποψήφια για δύο διαφορετικά πόστα. Πραγματικά θα ήθελα ο κανόνα σα, ο κανόνα στον οποίο να αναφερθήκατε, να μην ισχύσει αύριο. Για έναν πολύ απλό λόγο. Θα ήθελα να μην είμαι μόνη. Να μην είμαι μόνη στο ε, Governing Council τη ΕΚΤ, διότι αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα θα μείνω σαν καλαμιά στον κάμπο ε, για πολύ καιρό. Η κυρία Φόντερ Λάιεν λοιπόν είπε ότι μπορεί να εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας και εγώ είμαι πραγματικά ένθερμη υποστηρίκτρια της ίσης εκπροσώπησης των φίλων. Αύριο λοιπόν μια καλή εξισορρόπηση ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως στοιχείο που θα φροντίσει να έχουμε άλλη μια γυναίκα στο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΕΚΤ. Μην το πάρετε πολιτικά το σχόλιο, αλλά πραγματικά το λέω για προσωπικούς λόγους. Θα θέλαμε να υπάρχει και στο Συμβούλιο Διευθυντών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ακόμα μία γυναίκα. Και αυτή η ίσα εκπροσώπηση. Τώρα, δεύτερο θέμα, οι κλιματικές αλλαγές. Το είχα πει και στην ακρόασή μου, μετά την οποία ψηφίστηκα και υπερψηφίστηκα. Είμαι πεπισμένη για την κέρια, την πρωταρχική σημασία της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει θα πρέπει να ε, διερευνήσει, να κοιτάξει και να μελετήσει πώς μπορεί καλύτερα να συνεισφέρει στην καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων των αλλαγών στο κλίμα. Δεν είναι βασική μα εντολή, βέβαια, το να ασχοληθούμε με την καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, αλλά είναι η σταθερότητα των τιμών. Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα έχει και μια εντολή που δεν είναι, ας πούμε, πρωτογενής, αλλά ως δευτερογενής εντολή και αρμοδιότητα, ε, είναι να υλοποιεί όλε τι αποφάσει που λαμβάνονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Έτσι, κατά συνέπεια, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι κλιματικέ αλλαγέ, οι επιπτώσεις τους είναι μέρος της εντολής μας, ε, τουλάχιστον δευτερογενός. Αυτό που ελπίζω είναι ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής αναθεώρησης που θα ξεκινήσει, τις ερχόμενες εβδομάδες, να μπορέσουμε και ελπίζω ότι αυτό πραγματικά θα βρει σύμφωνο και το Συμβούλιο των Διευθυντών, ε, ελπίζω να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε το στοιχείο των κλιματικών αλλαγών ως ε, αναπόσπαστο τμήμα για να δούμε πώς και σε τι βαθμό η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να το λάβει υπόψη. Ξέρω ότι είναι σημαντικό και για μένα είναι ιδιαίτερα προσφυλές και αν μου επιτρέπετε γι' αυτό να παρα... ξεπεράσω λίγο το όριο του χρονομιλία. Παράδειγμα, για τι προβλέψει ε, τι μακροοικονομικέ. Χρησιμοποιεί μοντέλα, μακροοικονομικά μοντέλα Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει, εξελαχίστων τουλάχιστον, τα μακροοικονομικά αυτά μοντέλα να ε, συμπεριλαμβάνουν στην εκτίμηση των κινδύνων που γίνεται του κινδύνου λόγω των κλιματικών αλλαγών. Το ελάχιστο μπορούμε να κάνουμε αυτό. Και κατά δεύτερον, στην ε, λειτουργία εποπτεία τη πρέπει η ΕΚΤ να μπορεί, χάρη σε δηλώσει, σε δεσμεύσει διαφάνεια στα πλαίσια εποπτεία των τραπεζικών ιδρυμάτων να καθορίζει κατά πόσον τα τραπεζικά ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη αυτέ ακριβώ τι κλιματικέ αλλαγέ όταν εκτιμούν του κινδύνου και ταυτόχρονα καθορίζουν το χαρακτήρα των ε, χρηματοπιστωτικών ε, προϊόντων. Και μετά για το σύστημα των συντάξεων της ΕΚΤ. Υπάρχει ήδη μια πολιτική που εφαρμόζεται για να δοθεί προτεραιότητα στα ε, χρηματοπιστωτικά εργαλεία τα οποία ονομάζονται πράσινα εντό εισαγωγικών. Και το βρίσκω απόλυτα θεμετό στα πλαίσια της εντολής μας. Και με ιδιαίτερη προσοχή στο να διατηρείται η οικονομική σταθερότητα βέβαια αμύωτη, νομίζω ότι καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κοιτάξει και τον τρόπο με τον οποίο οι ε, διάφορες συναλλαγές και όλες τις ενέργειες ε, διενεργούνται με ιδιαίτερη έμφαση στην συνεκτίμηση των κλιματικών αλλαγών. Ωραία. Και τώρα ο κύριος Γιούνας από τους Πρασίνους. Thank you, Chair. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να σας καλωσορίσω κυρία Πρόεδρε και επικροτώ τον ε, ανοιχτό τρόπο με τον οποίο εκφράζεστε και τις φιλοδοξίες σας θα δούμε στο μέλλον τα αποτελέσματα της φιλοδοξίας αυτής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το ψηφιακό νόμισμα της Κεντρικής ε, Τράπεζας, αλλά πρώτα θα ήθελα να αναφερθώ στην αναντιστοιχεία ε, ασφάλειας ε, και ρίσκου των στοιχείων του ενεργητικού. Ε, παραμένει θέμα το ότι οι τράπεζες είναι υπερβολικά συνδεδεμένες μεταξύ τους ε, για να τις αφήσουμε ε, να χρεοκοπήσουν. Υπάρχει ο ηθικός κίνδυνος, μας ενδιαφέρουν τα κίνητρα και επίσης πρόβλημα είναι τα κίνητρα για αύξηση του βραχυπρόθεσμου κέρδους. Έχουμε τα stable coins, έχουμε ε, τα εικονικά νομίσματα, όπως και να θέλετε να τα ονομάσετε, και αυτά αποτελούν ε, θέμα. Αναφερθήκατε στην αλλαγή του κλίματος, ε, την θεσμοθέτηση των τιμών κλπ. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν η εντολή για οικονομική σταθερότητα μπορεί να διευρυνθεί και να ε, συγκεκριμενοποιηθεί. Πώς βλέπετε τα ψηφιακά νομίσματα ως πιθανή λύση για τα προβλήματα αυτά. Ξέρω ότι μιλάτε από μια συγκεκριμένη γωνία, αλλά θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, για παράδειγμα, με την Ρίξπαν και ε, μέχρι πότε προβλέπετε να έχουμε αποτελέσματα σχετικά με αυτό το ψηφιακό νόμισμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ουσία της εντολής είναι η σταθερότητα των τιμών, όχι η οικονομική σταθερότητα. Τούτου λεχθέντος, ε, φυσικά μια κεντρική τράπεζα πρέπει να ε, αφουγκράζεται τις ε, οικονομικές εξελίξεις, ε, τις χρηματοοικονομικές εξελίξεις και την σταθερότητα του οικονομικού τομέα, καθώς και τις τάσεις στον βαθμό που επηρεάζουν την σταθερότητα των τιμών. Όσον αφορά το ψηφιακό νόμισμα της Κεντρικής Τράπεζας, προσπάθησα στην εισαγωγή μου να αναφερθώ σε δύο τομείς. Πρώτον, θα πρέπει να μπορούμε να αναλύουμε και να μετράμε τον αντίκτυπο ε, στην ε, οικονομική πολιτική ε, με όρους οικονομικής σταθερότητας. Και τα δύο αυτά έχουν μεγάλη σημασία, διότι εάν θέλουμε να αναπτύξουμε αυτό το ψηφιακό νόμισμα της Κεντρικής Τράπεζας, θα πρέπει να σκεφτεί κανείς καταρχάς την ασφάλεια, την ασφάλεια του καταναλωτή. Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα ε, και την ασφάλειά του, τον ρόλο που παίζουν οι εμπορικές τράπεζες και το πώς οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το νόμισμα. Ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα αυτά μαζί και ελπίζουμε αυτό να γίνει ενώ θα προχωράμε στην ψηφιοποίηση των νομισμάτων. Αυτό είναι ένα εγχείρημα που γίνεται σε διάφορα φόρουμ. Γνωρίζετε ότι το BIS ε, με τον ε, κόμβο καινοτομία ε, θα είναι ιδιαίτερα δραστήριο. Είναι κάτι που επίσης γίνεται σε άλλα επίπεδα. Θέλουμε να δούμε λοιπόν πώς η καινοτομία μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια και την αξιοπιστία του συστήματος. Ξέρω ότι και η Σουηδική Κεντρική Τράπεζα έχει ασχοληθεί ενεργά με την ανάπτυξη ψηφιακού νομίσματος της Κεντρικής Τράπεζας, όπως και η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας. Και η PBOC στη στην Κίνα προσπαθεί να αναπτύξει ένα παρόμοιο σύστημα. Πιστεύω ότι είναι ένας τομέας όπου θα πρέπει να σπέβδουμε βραδέως, διότι φυσικά υπάρχει ζήτηση, είναι μια τεχνολογία αναπτυσσόμενη που θα μπορέσει να στηρίξει μια τέτοια καινοτομία, αλλά όταν λέω ε, βραδέως ε, πρέπει να γνωρίζουμε τους κινδύνους ε, που θα κινητοποιήσει ένα τέτοιο σύστημα και όσον αφορά το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα και το οικονομικό σύστημα στο σύνολό του. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ελέν Λαπόρτ από το ID, παρακαλώ. Κύριε Λαγκάρτ, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για την ανταλλαγή αυτή. Τελευταία, έχετε πει ποια θα είναι τα κεντρικά σημεία της νομισματικής ε, πολιτικής. Είσαστε στη θέση σας από τον Νοέμβριο. Σε συνέχεια, με τον κύριο Ντράκη είπατε ότι είσαστε υπέρ της διευκολυντικής αυτής νομισματικής πολιτικής, ότι είσαστε υπέρ των χαμηλών ε, επιτοκίων και της ποσοτικής χαλάρωσης. Και όλα αυτά με τριπλό στόχο, απόλυτα θεμητό, να αντιμετωπιστεί ο αποπληθωρισμός, ο ανάπτυξη της οικονομίας κατά της ανεργίας. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με το ίδιο το καθεστώς της ΕΚΤ που έχει σαν στόχο ε, μοναδικό την σταθερότητα των τιμών και τον πληθωρισμό στο 2 ή Πρέπει όμως να δούμε το θέμα της παραγωγικότητας, το θέμα της απασχόλησης. Η ΕΚΤ αυτό τον κανόνα, τον χρυσό που την εμποδίζει να χρησιμοποιήσει ένα σωρό άλλα του που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πόσο πολύ τον θέλετε και δεν θα μπορούσε να έχει μια νομισματική πολιτική αντικυκλική ε, αν δεν είχε τόσο περιορισμένα περιθώρια λιγμών. Δεν θα ήταν καλύτερα να είναι ο πληθωρισμός 1% το χρόνο και να μπει στο καθεστώς της ΕΚΤ και άλλα στοιχεία πέρα από αυτά που έχει τώρα. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός προπολογισμού της Ευρωζώνης. Κάτι το οποίο στηρίξατε εσείς με τον πρόεδρο Μακρόν, αλλά δεν πέτυχε υποστήριξη από πολλούς. Η δημιουργία ενός προπολογισμού στην Ευρωζώνη σημαίνει ότι θα διευκολυνθούν και οι μεταφορές μεταξύ των χωρών ε, μελών. Με τι ποσό όμως και ποιο θα είναι το κόστο της Γαλλίας που ήδη είναι καθαρός εισφορέας ε, με ήδη 8 δισεκατομμύρια το 2018. Πώς θα διαρθρωθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την, ερωτήση, την ερώτησή σας. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω στα αγγλικά, λέει κυρία Λαγκάρτ. Πρέπει να έχω κι εγώ μια καλή ισορροπία. Ε? Πριν μίλησα για πολύ στα γαλλικά. Λοιπόν, αγγλικά. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό θα είναι και το εγχείρημα που θα ακολουθήσουμε στα πλαίσια της αναθεώρησης της στρατηγικής μας. Δηλαδή, θα αναρωτηθούμε. Το 2003 Αυτά αποφασίστηκαν. Κοντά ή κάτω από το 2%. Με όλες τις αλλαγές που έχουν λάβει η χώρα, τις οικονομικές συνθήκες, τις τάσεις που παρατηρούμε, θα εξετάσουμε κατά πόσο αυτός ο ορισμός της σταθερότητας των τιμών και αυτή η στόχη που είναι της ΕΚΤΑ, και που πλαισιώνουν τη σταθερότητα τιμών, θα δούμε κατά πόσο εξακολουθούν να ισχύουν, σε τι βαθμό, ε, με ποιο τρόπο, με τι περιθώρια. Ε, είναι ένας ε, στόχος, είναι μια προσπάθεια. Θα υπάρξουν πολλές αποχρώσεις που θα συζητηθούν στα πλαίσια του στόχου μας για τον πληθωρισμό που θα συζητηθούν. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα δεν το γνωρίζουμε φυσικά σε αυτό το στάδιο. Πάντως θα πρέπει να αναποδογυρίσουμε κάθε πέτρα, θα πρέπει να εξετάσουμε κάθε εναλλακτική και όπως είπα και νωρίτερα στις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις θα είναι μία ανάλυση σε βάθος και με ανοιχτό το πνεύμα. Πάντως, στο τέλος, αυτό που μας νοιάζει είναι η εντολή της ΕΚΤ που είναι η σταθερότητα τιμών. Και έχει αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο που συνεισέφερε τα τελευταία χρόνια μάλιστα για την ε, σταθερότητα των τιμών και βοήθησε στην ανάπτυξη, στη δημιουργία απασχόλησης και κατά τη γνώμη μου η χρήση αυτής της πολιτικής και η χρήση των μέσων, των εργαλείων πάνω στα οποία βασίστηκε η ΕΚΤ ήταν αναγκαία και τα κατάλληλα προκειμένου να έχουμε τα αποτελέσματα που είχαμε. Τώρα για τη δεύτερη ερώτησή σας, ομολογώ ότι δεν ε, πολύ κατάλαβα τη δεύτερη ερώτησή σας. Ίσως θα μπορούσε να επαναλάβει το δεύτερο σκέλος. Ναι, είναι για τον προπολογισμό της Ευρωζώνης. Α, ναι, και ε, το έλεγα γιατί εμείς συνεισφέρουμε 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν με τι ποσό θα έπρεπε να συνεισφέρει η Γαλλία σε έναν τέτοιο κοινό προπολογισμό της Ευρωζώνης. Απάντηση. Δεν θα σας εκπλήσει η απάντησή μου. Στο βαθμό που υπάρχει μία νομισματική ένωση που είναι η Ευρωζώνη και έχει νόμισμα το ευρώ, θα ήταν ευπρόσδεκτο και θα μας έβαζε στην ίδια κατηγορία με άλλες νομισματικές ένωσεις, εάν είχαμε και μία οικονομική ικανότητα, τώρα αν θα ήταν μεγάλη, ε, ξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα, τη σύγκληση ή αν ακόμα καλύτερα θα συμπεριλαμβάνει και ένα στοιχείο σταθερότητας, αυτό θα αποτελούσε μία βελτίωση στην όλη αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Χωσέ Κουσμάου τώρα. Γκουε, α, όχι. Α, συγγνώμη. Ο κύριο Όφερφελτ από το ECR, ζητώ συγγνώμη. Ο κύριο Φανόβερφελτ. Είμαι εδώ. Καλησπέρα σα Εδώ είμαι. Ευχαριστούμε που είστε εδώ, κύριε Λαγκάρντ. Έχω τρει ερωτήσει για εσά. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Πρώτα απ' όλα για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών είναι μια κρίσιμη προτεραιότητα για την ΕΚΤ ε, θεωρητικά. Αλλά ταυτόχρονα ο κύριος Βάιτμαν από την ε, Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Γερμανίας λέει ότι η νομισματική πολιτική που θα επιδιώκει ρητός περιβαλλοντικούς στόχους μπορεί να ε, δημιουργήσει πρόβλημα. Ήθελα σχόλιο για την δήλωση Whiteman και μετά για τις κρατικές επενδύσεις. Είπατε ότι είστε υπέρ Είπατε τέλο πάντων ότι χρειάζονται περισσότερε δημόσιε επενδύσει. Δύο υπερωτήσει λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θα υποστηρίζετε μια πρωτοβουλία για την εξαγορά ελλείμματο ε, και αυτό που έκριναν οι ευρωπαϊκέ ε, αρχέ ότι το 3% έλλειμμα θα πρέπει να μην λαμβάνει υπόψη το ποσοστό των επενδύσεων και μετά πώ πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει δημόσια χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων. Και μετά Είπατε για την παραγωγικότητα ότι πρέπει να βελτιωθεί, το δηλώσατε πρόσφατα, όμω βλέπουμε τα χαμηλά επιτόκια για τι τράπεζε. Αυτά οδηγούν σε επιβράδυνση τη παραγωγικότητα με ε, την διατήρηση στη ζωή των λεγόμενων εταιριών και επιχειρήσεων ζόμπι. Παρακαλώ σχολιάστε το. Μάλιστα, ε, ευχαριστώ για τις κλιματικές αλλαγές. Όπως είπα, στην προηγούμενα σχολεία μου, Ως κεντρική τράπεζα πρέπει να διερευνήσουμε όλες τις παραμέτρους της δουλειάς μας, αυτές που οργανώνουμε, στις οποίες λειτουργούμε και τις ενέργειες που φέρνουμε εις πέρας. Οι κλιματικές αλλαγές λοιπόν είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο, πρέπει να δούμε πώς θα ε, συμμετάσχουμε στον αγώνα της καταπολέμησής του. Αυτό εδώ συμφωνώ με τον κύριο Βάιτμαν. Δεν σημαίνει ότι η πρώτη μα αρμοδιότητα είναι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Δεν είναι δική μα αποστολή. Οι κυβερνήσει, οι πολιτικοί ηθήνοντε, εκείνοι πρέπει να καταδιδραματίσουν τον πρωταρχικό ρόλο. Δεν μα εμποδίζει όμω από το να κοιτάξουμε τη δική μας λειτουργία και να δούμε όλες τις συνιστώσεις για να είμαστε αποτελεσματικότεροι. Όπως είπα προηγουμένως, δυστυχώς ίσως στα γαλλικά, αλλά το πω και στα αγγλικά, πρώτον, στην μακροοικονομική μας ανάλυση πρέπει να συμπεριλάβουμε στην δημιουργία μοντέλων, μακροοικονομικών μοντέλων που είναι από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε, τι κλιματικέ αλλαγέ. Πρέπει να συμπεριληφθούν εκεί. Μετά, στην εποπτεία, την επιθεώρηση των τραπεζών, πρέπει να συμπεριληφθούν οι κλιματικέ αλλαγέ. Βεβαίω, στη διακυβέρνηση τη Κεντρική Τράπεζα και του Ευρωσυστήματο υπάρχουν φορέ που το απαιτούν. διαφάνεια το απόρριτο και η δημοσιοποίηση, η αξιολόγηση του κινδύνου πρέπει να είναι τμήμα της εποπτείας που διεξάγουν οι εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του SSM. Και τρίτον, πρέπει να συμπεριλάβουμε τις κλιματικές αλλαγές και τις επιταγές τους, τις ε, ε, συναλλαγές, τις επενδυτικές, αυτές που φέρνουμε εις για το δικό μας το χαρτοφυλάκιο και για την διαχείριση των συνταξιδοτικών ταμείων. Αυτά τα κάνουμε ήδη, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Για να δούμε πόσα μπορούμε να κάνουμε. Και στο πρόγραμμα αγορών μας πρέπει να δούμε πόσο οι κλιματικές αλλαγές έχουν κάποιον αντίκτυπο. Γι' αυτό θα το καθορίσει αυτό έτσι καλλιώ το Συμβούλιο των Διευθυντών, το Διοικητικό Συμβούλιο τη Τράπεζα. Εκεί θα γίνουν συγκεκριμένε προτάσει και θα συζητηθούν για να ληφθούν αποφάσει. Όμω αυτοί οι τέσσερι τομεί μου φαίνονται σημαντικοί και εκεί έχουν ε, επίπτωση κλιματικέ αλλαγέ. Με ρωτήσατε για τι επενδύσει. Δεν είναι η δική μου δουλειά να δω τι εξονυχιστικέ λεπτομέρειε για το τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τι όχι το έλλειμμα το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη, το Δίπτυχο και το Εξάπτυχο που θα αναθεωρηθούν, ε, τα διευκρινίζουν αυτά και εκεί θα πρέπει να απαντηθούν οι ερωτήσει σας. Από τη δική μου τώρα την σκοπιά και από τη σκοπιά της σταθεροποίηση των τιμών χρειαζόμαστε βεβαιότητα και ασφάλεια. Χρειαζόμαστε σαφήνεια. Νομίζω λοιπόν και είναι κοινή άποψη στην κοινότητα των οικονομολόγων και των εμπειρογνωμόνων στα θέματα αυτά, ότι τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ιδιαίτερα περίπλοκα. Κάποιε φορέ η σκοπή είναι αλληλένδεται ανάλογα με το πώ θα ορίσει κανεί το κάθε θέμα, οπότε αν βρούμε έναν τρόπο να τα ορίσουμε σωστά, σίγουρα θα προχωρήσουμε και απλούστερα προ τον σκοπό μα. Απαντώντας την πρώτη ερώτηση, ε, εξέφρασα μια ανησυχία για το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων εν γέννη, όχι μόνο για τις κρατικές επενδύσεις. Δεν είμαι βέβαια ότι η ΕΚΤ μπορεί εδώ να αναλάβει σημαντικό ρόλο για συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων. Ε, πρέπει βεβαίως να προσφέρουμε χρηματοδότηση με κόστος ε, ελκυστικό, ώστε και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να ενθαρρυνθούν για να κάνουν κάτι προ αυτή την κατεύθυνση. Και ρωτήσατε και για την παραγωγικότητα. Η επένδυση στην καινοτομία, στην τεχνολογία και την ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη της οικονομίας, αυτό θα οδηγήσει σε βελτίωση της παραγωγικότητας. Και χρειαζόμαστε επενδύσει για να μπορέσει η οικονομία μας να είναι παραγωγικότερη. Ευχαριστώ. Now... Σα ευχαριστώ πολύ. Μανομπρία από την ΚΟΕ. Euh, Καλημέρα κύριε Λαγκάρτ. Θα συνεχίσω στο βασικό θέμα που κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι η προτεραιότητα, αλλά τέλος πάντων μια προτεραιότητα, εσείς άλλο το λέτε προτεραιότητα άλλο μια μεγάλη προτεραιότητα, το κλίμα. Εδώ έχω το κείμενο των 160 μη κυβερνητικών οργανώσεων. Το βήμα αυτό και ο λόγος των πολιτών είναι κάτι για το οποίο θα ήθελα να σας ενημερώσω, γιατί ζητούν κάτι πολύ συγκεκριμένο και με ταχύτητα. Ακούγοντας αυτά που λέτε, βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέτε ότι θέλετε να ασχοληθεί με το κλίμα και πράγματι όλες οι δηλώσεις που έχετε κάνει είναι θετικές και σας ενθαρρύνουμε. Λέτε ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι στην καρδιά της ΕΚΤ κλπ. κλπ. Συμφωνούμε. Τώρα, πώς θα περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις. Πρώτον, η ΕΚΤ. Ξέρουμε ότι και αυτή συνεισφέρει με δισεκατομμύρια που έχει επενδύσει στα ορυκτά καύσινα και σε πολυεθνικές όπως η Σέλιπη κλπ. Και συνεχίζει να το κάνει και θα συνεχίσει όταν το μόνο που την απασχολεί είναι η ουδετερότητα των αγορών. Σήμερα μας είπατε ότι θα υπάρξει αναθεώρηση της στρατηγικής Τη νομισματική τη ΕΚΤΕ που δεν έχει αλλάξει από το 2003 όπω είπατε. Αλλά μήπω θα μπορούσατε να μα πείτε περισσότερα για το χρονοδιάγραμμα. Πότε θα γίνουν όλα αυτά. Πώς θα συμπεριληφθεί η κλιματική αλλαγή. Και ένα άλλο ζήτημα είναι πώς χρηματοδοτούμε πράσινες επενδύσεις και πώς βγαίνουμε από τις καφέ, τις βρώμικες επενδύσεις όπως το ζητάει η κοινωνία των πολιτών, που ζητάει από τώρα η ΕΚΤ να αποποιηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στα ορυκτά. Μπορείτε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα πώς θα το πετύχετε αυτό. Και χωρίς να περιμένουμε την ε, ταξινόμηση που ξέρουμε ότι θα πάρει χρόνο γιατί συμμετέχει και το Συμβούλιο σε αυτήν. Η κυρία Λαγκάρτ. Ευχαριστώ, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θα διαφωνήσω μαζί σας στο τελευταίο. Γιατί όλοι είμαστε μαζί στο ίδιο καράβι για αυτά. Δεν μπορούμε να πούμε, α, εσύ θα κάνεις αυτή τη δουλειά, εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, η ταξινόμηση θα έρθει όταν έρθει. Όχι. Είναι ζωτική σημασία να την έχουμε γρήγορα την ταξινόμηση αυτή. Και δεν θέλω βέβαια να παρέμβω εδώ και να αναμειχθώ στις δικές σας συζητήσεις γιατί δεν, είναι, δεν είμαι και η κατάλληλη, αλλά ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει αυτή η ταξινόμηση και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία προχωρώντας τις δράσεις μας. Τώρα, σίγουρα θα υπάρξουν διαφωνίες, μετάβαση με μετάβαση, πώς, ε, πόσο ε, λεπτομερώς θα εξετάσουμε το τι γίνεται και το τι κάνουμε και τι είναι ακριβώς αυτές οι επενδύσεις. Πάντως ελπίζω να υπάρξει πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά κάποιο τρόπο είναι κάτι σημαντικό. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, προσπαθώ να εντοπίσω σε ποιους τομείς κατά τη, γνώμη μου δηλαδή και έχοντας υπόψη ότι μόνο τέσσερις εβδομάδες είμαι στο έκτα, πιστεύω ότι μπορεί να επηρεάσει. Στον εντοπισμό καταρχήν στην μακροοικονομική ανάλυση όπου θα λάβουμε υπόψη μας την κλιματική αλλαγή. Όταν ε, φτιάχνουμε και διαμορφώνουμε μοντέλα, όταν κάνουμε προβλέψεις, όταν προσπαθούμε να εντοπίσουμε και να προβλέψουμε αναμενόμενο πληθωρισμό κτλ. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τη συμπεριφορά των οικοκυριών. Γιατί αγοράζουν αυτό και όχι το άλλο. Ε, γιατί ψωνίζουν εκεί και όχι αλλού. Γιατί παίρνουν σπίτι Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και να ενσωματώσουμε την κλιματική διάσταση ε, σε όλη αυτή την ανάλυση που κάνουμε. Κάτι το οποίο σίγουρα χρειάζεται χρόνο και κόπο, αλλά θα γίνει. Και ελπίζω να υπάρξει συμφωνία από όλες τις πλευρές. Είναι κάτι το οποίο το θέλω. Θα υπάρξει όμως απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο σε διάλογο μαζί σας και την κοινωνία των πολιτών. Μισή ώρα ήμουνα πριν με αυτούς ακριβώς που έχουν υπογράψει το κείμενο που μου δείξατε. Και θέλω να συνεχιστεί ο διάλογος. Τους χρειάζομαι. Χρειάζομαι να καταλάβω κι εγώ τον τρόπο που εκείνοι ε, προσεγγίζουν το ζήτημα. Τώρα, το άλλο σημαντικό βέβαια είναι η εποπτεία. Αυτό αποτελεί ένα σκέλος, ένα μέσο που διαθέτει η ΕΚΤ και μπορεί να το χρησιμοποιήσει για καλό σκοπό. Οι ε, διοικητές των κεντρικών ε, τραπεζών και οι υποπτικές αρχές των χωρών μελών επίσης πρέπει να κάνουν το δικό τους, τη δικιά τους δουλειά. Ε, για τις άμεσες επενδύσεις, για παράδειγμα, όπως είπα και πριν, όπου έχουμε πολλά προϊόντα τα οποία ονομάζονται πράσινα, παρόλο που δεν είναι ακόμα έτοιμη η ταξινόμηση. Όσον αφορά τώρα για το πρόγραμμα αγορών, 80% ε, των αποθεμάτων των προϊόντων που έχουμε είναι κυβερνητικά ομόλογα και είμαστε ένας από τους κύριους αγοραστές των ομολόγων που εκδίδουν διεθνείς οργανισμοί στην Ευρώπη που δεσμεύονται να επενδύουν μόνο σε πράσινες επενδύσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τώρα υπάρχει και ένα μικρό ιδιωτικό κομμάτι, όπου εκεί υπάρχουν ε, διάφορες αποχρώσεις από το πράσινο μέχρι το καφέ. αλλά πρέπει να προσέξουμε ε, να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στην ε, αγορά ξαφνικά και να τηρήσουμε βέβαια και την αρχή της ουδετερότητας η οποία εφαρμόζεται. Πρέπει να αναθεωρηθεί με ποιο τρόπο αυτό ακριβώς θα αποτελέσει μέρος της αναθεώρησης της στρατηγικής μας, της συζήτησης δηλαδή που θα κάνουμε για την αναθεώρηση της νομισματικής μας στρατηγικής. Σας ευχαριστώ κύριο Σενίντερ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, χαιρόμαστε που βρίσκεστε εδώ. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με την οικονομία και την νομισματική πολιτική. Είπατε στην αρχική σας εισήγηση ότι η οικονομία είναι αρκετά εύθραυστη, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έλαβε σοβαρά μέτρα για υποστήριξη της οικονομίας. Πιστεύετε ότι στο μέλλον θα μπορέσετε να κινητοποιήσετε περαιτέρω την ε, οικονομία για να μην ολιστήσουμε ε, σε στασιμότητα ή ύφεση. Ε, εκτιμώ την προσήλωσή σας ε, στα διάφορα θέματα που αναφέρατε, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω ε, νομισματικά σύνολα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο παρελθόν θα συνεχίσουν να παίζουν τέτοιο ρόλο, διότι πολλές κεντρικές τράπεζες είναι πολύ σκεπτικές όσον αφορά αυτά τα μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, η οικονομία θα μπορούσε να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και πράγματι είπα ότι κυρίως σε εξωτερικούς παράγοντες οφείλεται η αργή ανάπτυξη ε, και σίγουρα βρίσκεται πιο χαμηλά από τις δυνατότητες. Έχουμε ε, τα, τα εργαλεία να αντιδράσουμε, ε, ναι, τα έχουμε και είμαστε αποφασισμένοι να τα χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί. Όπως σας είπα, η εντολή μας είναι η σταθερότητα των τιμών και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι απαιτείται. Φυσικά όλοι οι διάφοροι παράγοντες ε, θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους ε, όσον αφορά τα monetary aggregates. Ε, είναι δύσκολο να προβλέψουμε τι θα κάνουμε όσον αφορά τη στρατηγική αναθεώρηση. Ε, όσον αφορά λοιπόν ε, τα νομισματικά μεγέθη, ε, δεν γνωρίζω ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, αλλά θα βλέπουμε ότι οι κεντρικές τράπεζες αρχίζουν να έχουν κάποιο αντίκτυπο και ανάλογα με την δημιουργία νέου χρήματος, είναι μια θεωρία που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ, ο Πολ Τάγκ από το S&D. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Αλαγκάρτ επικροτώ τα λόγια σας σχετικά με το πώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να ενσωματώσει μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη ε, την αλλαγή του κλίματος ε, εντός ε, της εντολής της για σταθερότητα των τιμών. Αυτό ακούγεται πολύ ενθαρρυντικά. Μερικές φορές όμως θα ήθελα πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο προκατοχός σας, ο Μαριο Ντράγκη, είπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ότι σχετικά με το CSPP ότι θα ε, το εξετάσει το θέμα ε, όσον αφορά δηλαδή το οικολογικό αποτύπωμα. Έχει γίνει μια τέτοια αξιολόγηση. Εάν ναι, μπορείτε να μας δημοσιεύσετε τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης. Ε, πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική δημοσίευση της, του οικολογικού αποτυπώματος όσον αφορά την ταξινόμηση. Το δίκτυο για το πρασίνισμα, τον οικολογικό προσανατολισμό του οικονομικού συστήματος ε, ε, έχει δώσει μια σύσταση ότι χρειαζόμαστε μια σαφή ταξινόμηση πράσινων ε, καφέ και άλλων προϊόντων. Συμφωνείτε με τη σύσταση αυτή του NGFS για γενική ταξινόμηση, όχι μόνο για τα πράσινα και καφέ προϊόντα, αλλά τις διάφορες αποχρώσεις τους. Τέλος, η κυρία Φοντερ Λάιεν είπε ότι ε, δεν ε, θα επιτρέψει ε, τον οικολογικό προσανατολισμό να να επιτρέψει δημοσιονομικά έλλειμματα. Πιστεύετε ότι αυτό το greenwashing αποτελεί κίνδυνο και πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξει αυξημένη κρατική δαπάνη για να γίνουν οι οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο βιώσιμες. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας ε, διαβάσω μια, ε, ένα έγγραφο το οποίο όμως είναι πριν από την εποχή μου. Θα ήθελα όμως να καταλάβετε ότι πράγματι η προσήλωση του κυρίου Ντράγη έγινε πραγματικότητα. Είχε δεσμευτεί να εξετάσει ε, το CSPP και έγινε μια προκαταρχική έρευνα και συνεχίζονται οι εργασίες. Για παράδειγμα, εξετάσαμε τις αγορές μας σε CSPP και διαπιστώσαμε ότι έχουμε αγοράσει πολλές πολλά πράσινα ομόλογα. Επίσης, σε άρθρο του 2018 λέει ότι το ευρωσύστημα ε, έχει δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τα πράσινα ομόλογα και υποστήριξε την ε, έκδοσή τους. Διαποστήσαμε όμως ότι ε, όσον αφορά το οικολογικό αποτύπωμα ολόκληρων οικονομικών τομέων, ε, όπως έχει γίνει από κάποιο Ινστιτούτο, μπορεί να είναι παραπλανητική. αγνοείται η δυναμική εντός των διαφόρων επιχειρήσεων σε βάθος χρόνου, το οποίο σημαίνει ότι αυτέ οι αναλύσει δίνουν ε, ε, ε, ημιτελή εικόνα, μη πλήρη εικόνα. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε το μέλλον, θα πρέπει να δούμε τι επενδύσεις χρηματοδοτούνται από κάθε επιχείρηση. και νομίζω ότι πίσω από αυτό το τελευταίο, πτώση, η έρευνα έγινε, μπορείτε να ε, την διαβάσετε και να διαβάσετε τα συμπεράσματα της συγκεκριμένη ε, μελέτης ε, που έδειξε ότι ο τρόπος χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ενθαρρύνει την έκδοση πράσινων ομολόγων. Ο πρόεδρος Τράγη δεσμεύτηκε και πράγματι κατέληξε σε κάποιο συμπέρασμα. Αλλά αυτό που προσπαθώ να πω εδώ είναι ότι για να το αναλύσετε αυτό θα πρέπει να το κάνετε ε, με πολύ αναλυτικό τρόπο. Θα πρέπει να ε, εξετάσει όλους τους παράγοντες ε, κανείς και να διαπιστώσει τι επενδύσεις γίνονται και ενθαρρύνονται με υποσυγκεκριμένες συνθήκες. Δεν θέλω να κατονομάσω κανέναν, αλλά Μπορεί μια οντότητα ε, που εσείς θεωρείτε καφέ να επενδύσει σε ένα πολύ πράσινο πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν ε, πώς το βλέπετε, γι' αυτό θα πρέπει να είναι πολύ αναλυτική εξέταση. Αλλά αυτό είναι θέμα που θα συζητάτε εσείς. Πώς ε, συνδέεται η χρηματοδότηση με τη μετάβαση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τεράστιες ανάγκες χρηματοδότησης για να βοηθηθούν οι καφέ οντότητες να ε, γίνουν λιγότερο καφέ και περισσότερο πράσινες. Οι δαπάνες αυτές πώς μπορούν να εντοπιστούν και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε παρέχοντας χρηματοδότηση χαμηλού κόστους για να τους διευκολύνουμε στη μετάβαση αυτή. Είναι ε, δύσκολο να γίνουν οι μετρήσεις, είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πόσο αναλυτική θα πρέπει να είναι η ανάλυση για να είναι σωστή. Ε, θα το εξετάσουμε το θέμα και εσείς φυσικά θα συνεχίσετε ε, δικαίως να ρωτάτε σχετικά με το θέμα αυτό. Ε, πρόεδρος, ε, σας ευχαριστώ. Πρωτού προχωρήσουμε να σας ζητήσω μια χάρη, διότι ε, έχουμε ακόμα δέκα συναδέλφους που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Σας παρακαλώ λοιπόν να περιοριστείτε στη μία ερώτηση ο καθένας, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις ε, στην κυρία Λαγκάρτ. Ο κύριος Κέλεχερ από το Ρενιού. Ευχαριστώ πολύ και καλώ ήρθατε κυρία Λαγκάρτ. Πολύ σύντομα αναφέρεστε σε στρατηγική αναθεώρηση της ΕΚΤ. Από πλευρά τη αναθεώρηση αυτή καθ' και την ικανότητα ανάλυση των πολιτικών τη ΕΚΤ ε, και πρόβλεψη για την οργάνωση στο μέλλον και πολιτικές που θα ακολουθούν στο μέλλον, εσείς θα κοιτάξετε πολύ στενά στα πλαίσια της σημερινής σας εντολής, που είναι το κοντά αλλά κάτω από το 2% ή και πέρα από την εντολή σας, δηλαδή θα εξετάσετε και γενικότερα οικονομικά στοιχεία, οικονομική ανάπτυξη, επενδύσεις, την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδοτήσει την αποκαθροποίηση της ε, Ευρώπης, ε, τις ιδιωτικές επενδύσεις ή θα περιοριστείτε πολύ στην αναθεώρηση αυτή. Και θα υπάρξει μια ανεξάρτητη ανάλυση Λαμβάνοντα υπόψη την προηγούμενη αναθεώρηση που έγινε το 2003 και δεδομένου ότι ήσασταν επικεφαλή του Δούνου ε, γνωρίζετε τι πέρασαν οι διάφορε χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς υπέφεραν. Πιστεύετε ότι τώρα δεν θα ήταν η στιγμή να κοιτάξουμε και πέρα από την εντολή αυτή να κοιτάξουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και πώς μπορεί να τοποθετηθεί στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, έχουμε αργή ανάπτυξη, οι οικονομίες μας ε, υποφέρουν, μιλάτε για μεγαλύτερη παραγωγή, περισσότερο πρασίνισμα, αλλά όλα αυτά χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις. Οπότε να ρωτιέμαι, αυτές οι αδύναμες οικονομίες που έχουμε στην Ευρώπη, πού θα τις βρούνε αυτές τις επενδύσεις. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα. Και κυρίως για αυτό το πρώτο κανόνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για την ενίσχυση του ρόλου του ευρώ διεθνώς. Μπορείτε να μου απαντήσετε κατά πόσο θα αποτελέσει και αυτό μέρος της ε, αναθεώρησης της στρατηγικής σας. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, μου βάζετε πολλές και δύσκολες ερωτήσεις που ξεπερνούν τι κάνει... Να, δύο λεπτά μου λέει ο πρόεδρο, Ξεπερνάει λοιπόν την εντολή και τι αρμοδιότητες τη ΕΚΤ. Να διευκρινίσω ένα πράγμα. Η εντολή έτσι όπως εγγράφεται στη βασική μας νομοθεσία είναι η σταθερότητα των τιμών. Και σε αντίθεση με άλλα όργανα, εμείς έχουμε μία ενιαία εντολή. Η ΦΕΝΤΕ δεν έχει ενιαία εντολή, έχει τη σταθερότητα τιμών, αλλά έχει και την απασχόληση ως ε, εντολή, μέρος εντολής της. Τώρα, η σταθερότητα τιμών ορίστηκε το 2003 με το κοντά αλλά κάτω από το 2%. Και αυτός είναι ο στόχος μας που συμμορφώνεται με την εντολή μας που είναι η σταθερότητα τιμών. Συνεπώς, πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Να οργανώσουμε καλά την αναθεώρησή μας. Να δούμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε για να συμμορφωθούμε προς την εντολή μας. Τώρα, σίγουρα υπάρχουν και άλλες πτυχές πέρα από το στόχο του πληθωρισμού που θα έπρεπε να λυθούν υπόψη για να είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε προς την εντολή μας και συζητήσαμε για παράδειγμα το θέμα της κλιματικής αλλαγής και το πώς επηρεάζει και πού επηρεάζει την εντολή μας για σταθερότητα τιμών και πώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε κάθε βήμα και να συμπεριληφθεί τελικά στο έργο μας. Τώρα πρέπει να πάμε πολύ πιο μακριά από αυτό. Πρέπει να συμπεριλάβουμε στην αναθεώρησή μας και όλες τις άλλες πτυχές των ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών, τα δημοσιονομικά της Ευρώπης. Δεν νομίζω ότι αυτά θα αποτελέσουν τον πυρήνα της αναθεώρησης. Αν επηρεάζουν, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Ξέρετε όμως ότι η νομισματική πολιτική είναι περισσότερο αποτελεσματική και μπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσματα όταν συμπληρώνεται από άλλες πολιτικές. Τη δημοσιονομική, για παράδειγμα, πολιτική, από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να υπάρξει μετακύληση της νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία και στήριξή της. Αλλά δεν είναι αυτός σκοπός, δεν είναι ο πυρήνας της στρατηγικής της ΕΚΤ να ασχοληθεί με αυτά τα άλλα ζητήματα. Ευχαριστούμε και τώρα κυρία Χούμπνερ από το ΕΛΚ. Πραγματικά πολύ δυστυχής είμαι που πρέπει να περιοριστώ σε ένα μόνο ερώτημα, αλλά θα το κάνω, πρέπει να δώσω το παράδειγμα και στους υπολείπους. Ε, κυρία Λαγκάρτ, ε, Χθε είδαμε σε φωτογραφίε σα και την κυρία Φόντερ Λάιεν μαζί 50% ε, τη ευρωπαϊκή ηγεσία και πραγματικά αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Όμω ο κύριο Ντράκη, όταν έρχονταν εδώ στι περισσότερε ομιλίε του στο σώμα μα, τόνιζε ότι η ΕΚΤ έχει το βάρος εδώ και μια δεκαετία για την τόνωση της οικονομίας. Ε, και πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν ήταν ε, πολύ επιτυχημένος στο να περάσει την ιδέα για αυτή την ευθύνη και σε άλλου πολιτικού ευθυνόντε αυτού που ασχολούνται με τη δημοσιονομική κυρίω, ε, τη χάραξη τη δημοσιονομική πολιτική. Εσεί λοιπόν πώ το βλέπετε αυτό τα επόμενα χρόνια, θα συνεχίσετε την ίδια τακτική με τη δημοσιονομική πολιτική ή θα αρχίσετε να συμπληρώνετε τα τη δημοσιονομική πολιτική. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά χθε ήταν πολύ ευχάριστο υπήρχε πραγματικά μια αίσθηση ισότητας και ισοτιμίας με την πρόεδρο Φόντερ Λάιεν. Και μαζί και με τον πρόεδρο Σασόλη από κοντά. Τώρα για το συνδυασμένο αντίκτυπο που θα μπορούσαμε να έχουμε μαζί με την δημοσιονομική πολιτική θα ήταν πραγματικά πολύ ε, καλό και άλλες, παρα, οι άλλες του πολιτικού μείγματος να συνδυάζονταν για να αντιμετωπίσουμε την επιβράδυνση στην ανάπτυξη, αυτή την σπαζοκεφαλιά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Θα το κάνω και στο μέλλον, όπως έκανα και στο παρελθόν, αλλά πραγματικά πρέπει να κοιτάξουμε τα εργαλεία δημοσιονομικής πολιτικής που διαθέτουμε, τα οποία δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε εφόσον χρειάζονται. Πάντως, ε, οι άλλοι πολιτικοί θύνοντες πρέπει να παραδεχτούν πόσο σημαντικά είναι, μαζί με τη μόχλευση της δημοσιονομικής πολιτικής που θα υιοθετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε ότι τα επόμενα μέλη θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της κυρίας Χούμπνερ. Σας ευχαριστώ όντω. Ο λόγος στον κύριο Σούστερ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ε, πιστεύω ότι μπορώ να συντομεύσω, θα τα πω γερμανικά. Θα το πω όσο πιο σύντομα γίνεται, διότι ήδη δόθηκαν πολλές απαντήσεις που αφορούσαν το θέμα μου. Για το θέμα του κατά πόσον είναι αποτελεσματική πολιτική της ΕΚΤ, διότι τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλά για να αναχαιτιστεί ο πληθωρισμός, για να υπάρξει τόνωση λόγω της οικονομικής συγκαιρίας, αλλά δεν ε, τα καταφέραμε ακριβώς. Δεν πετύχαμε να ε, δώσουμε κίνητρα για επενδύσεις, για να ξεπεράσουμε τον πληθωρισμό του 1% που είναι πολύ χαμηλός και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την έκτα. Δεν είναι το πρόβλημα με τις επενδύσεις ότι, δεν είναι, ότι είναι χαμηλό το κόστος ε, και ότι δεν ε, μπορεί κανείς να λάβει τη χρηματοδότηση. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί πρώτον. Το βασικό πρόβλημα είναι το ίδιο το αρχιτεκτόνημα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Πρέπει δηλαδή να υποχρεωθούν όλοι να εργάζονται ταυτόχρονα. Όσοι σχεδιάζουν τον προπολογισμό με το δίπτυχο και το εξάπτυχο και τους περιορισμούς που προβλέπουν, πρέπει να κοιτάξουν με ε, τη συμμετοχή των διάφορων κυβερνήσεων, όπως ε, στη Γερμανία, με το στόχο αυτό των μηδενικών ποσοστών πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και πρέπει να δούμε από το 2003 όταν ξεκίνησε η Νομισματική και Οικονομική Ένωση τι συνεισφορά έδωσε η ΕΚΤ. Τι πρέπει να δούμε, ε, τι, πρέπει να τι μπορούμε να διορθώσουμε σε σχέση με αυτά που από τότε έχουν γίνει και ήταν επιτυχημένα. Ευχαριστώ. Μια μέρα ίσως να μπορώ να σας απαντήσω στα γερμανικά. Πρέπει να αναρωτηθεί κανείς είμαστε χρήσιμοι, συνεισφέρουμε σε κάτι για να το απαντήσουμε αυτό. Είναι και το με τι στόχο μετράει κανείς τις επιδόσεις του, δηλαδή κατά πόσον ο στόχος του και επετέχεται ή όχι. Ε, κοντά ή κάτω από το 2% ε, και δεν είμαστε ακόμα εκεί. Θα ήταν όμως ε, και σφάλμα να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι η ΕΚΤ δεν έχει κάνει και τίποτα διότι θα έπρεπε να δει κανείς το πράγμα και αντιστρόφως για να σκεφτεί αν κάναμε ότι μπορούσαμε ή αν πετύχαμε κάτι. Πρέπει κανείς να προσπαθήσει να καταλάβει τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε νομισματική πολιτική όπως αυτή που ακολουθήσαμε. Και θα βλέπατε ε, σε ένα τέτοιο σενάριο ότι ο αντίκτυπος στο επίπεδο του ΑΕΠ έχει ε, υπάρξει σημαντικός. 2,3 με 2,7% λένε τα μοντέλα των εκτιμήσεων. Το επίπεδο του ΑΕΠ θα ήταν χαμηλότερο αν δεν υπήρχε αυτή η νομισματική πολιτική. Το ίδιο για τον πληθωρισμό. Εάν δεν είχαμε αυτή την νομισματική πολιτική, ο πληθωρισμός θα ήταν ακόμη χαμηλότερος από ό,τι είναι σήμερα. ένα τρίτο ή μισή ποσοστία μονάδα. Όχι ότι είμαι πανευτυχής και θα πρέπει να είμαστε και ικανοποιημένοι με ό,τι κάνουμε. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμα καλύτερη δουλειά. Όλοι μας, όλοι οι πολιτικοί θύνοντες. Πιστεύω όμως ότι όντως η νομισματική πολιτική ήταν τόσο αποτελεσματική όσο μπορούσε τα τελευταία χρόνια. και το να έχουμε δημοσιονομική ικανότητα με το γνωστό ακρονίμιο που χρησιμοποιείται γι' αυτό, το εργαλείο σύγκλησης και ανταγωνιστικότητας, το να το έχουμε αυτό ως στοιχείο τη Νομισματική Ένωση, δημοσιονομική ικανότητα που να χρησιμοποιείται και για σκοπού σταθεροποίηση. Όταν μια χώρα αντιμετωπίζει ιδιαίτερου τρεγμού, θα πρέπει τότε να κοιτάξουμε και τους δεοντολογικούς κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν, αλλά και την προστασία μας από τα διάφορα ρίσκα. Δηλαδή θα πρέπει σίγουρα να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε την Μεσματική Ένωση. Ευχαριστούμε και τώρα κυρίως Γκίγκολτ από τους Πρασίνους. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ και χαίρομαι που τουλάχιστον υπάρχει μία γυναίκα στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ελπίζω σύντομα να έχουμε περισσότερες. Πέρα από αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και το τι μπορεί να κάνει η Κεντρική Τράπεζα. Όταν περιγράφατε τα συγκεκριμένα μέτρα που έχετε κατά νου, ήταν σαφές για μένα ότι ο πυρήνας της ε, νομισματικής πολιτικής δεν αναφέρθηκε. Δεν αναφέρθηκαν οι επιχειρήσεις αναχρηματοδότησης που είναι τόσο κρίσιμες. Ε, αυτές καθορίζονται από την αξιολόγηση κινδύνου. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, θα ασκήσετε πίεση στις, στους οργανισμούς αξιολόγησης ικανότητα ικανότητας ή στις δικές σας ε, αξιολογήσεις θα φροντίσετε στις ε, επιχειρήσεις αναχρηματοδότησής σας ε, να λαμβάνετε υπόψη η αλλαγή του κλίματος και όσον αφορά τις επιχειρήσεις ανοιχτής αγοράς όπως είναι η ποιοτική χαλάρωση, η ποσοτική χαλάρωση θα δώσετε τέλος σε ε, στις ανισορροπίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, διότι η αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα, έχει το 2,16% των ε, συνολικών ομολόγων, ε, ενώ στο δικό σας πρόγραμμα είναι 6,84%. Το ίδιο ισχύει για την ενέργεια, 2,55% συνολικά, ενώ πάνω από 9% για στο δικό σας ε, πρόγραμμα. Όλα αυτά είναι δεδομένα του 2017. Θα φροντίσετε λοιπόν να λαμβάνετε υπόψη ε, η αλλαγή του κλίματος και στον πυρήνα της ε, νομισματικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Καταρχάς, όσον αφορά την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, σίγουρα είναι ε, ζωτική σημασία όλοι οι οργανισμοί ε, να λάβουν υπόψη και τον ε, κίνδυνο αλλαγή του κλίματος. Αυτό δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε συγκεκριμένους οργανισμούς πιστοληπτικής ικανότητας και ελπίζω οι τρεις μεγάλοι οργανισμοί να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Και εάν ρωτήσουν την απόψή μου θα τους πω όπως ακριβώς το λέω και σε εσά αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, ε, τα προγράμματα αναχρηματοδότησης που έχουμε τώρα και που θα έχουμε στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν με βάση την ουδετερότητα της αγοράς ε, που έχει αμφισβητηθεί. Έχει λάβει διάφορες ερμηνείες από διάφορες πλευρές ε, και σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε ως μέρος της στρατηγικής και ως ε, τμήμα της αναθεώρησης ε, των εργαλείων που χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε το στόχο μας, ε, πρέπει να αναρωτηθούμε σχετικά με την καταλληλότητα, την αναλογικότητα και τη συμπερίληψη του κινδύνου αλλαγής του κλίματος στους παράγοντες. Ναι, πράγματι. Αλλά ναι, το προσέξατε κι εσείς. Όποτε μιλάμε για στρατηγική αναθεώρηση, Ε, προσέχω να μην ε, σας δώσω οριστική απάντηση, διότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πλαίσιο θα πρέπει να συμφωνηθεί από όλους και όχι. Ε, δεν είναι ατομική επιχείρηση, πρόκειται για συλλογική προσπάθεια και σε, διάλογο με εσά, με την κοινωνία των πολιτών και με εμπειρογνώμονες θα βελτιώσουμε το αποτέλεσμα. Και προσβλέπω σε αυτό. Ευχαριστούμε. Καρμπονάτο. ID παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ιταλικά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Λαγκάρτ που είστε εδώ. Πραγματικά εκτιμώ πολύ την ε, ανοιχτόμυαλη προσέγγισή σας σε σχέση με το αίτημα να αναθεωρηθούν οι στόχοι της ΕΚΤ. Ε, ε, το έθιξαν αρκετοί συνάδελφοι ως τώρα το ότι οι στόχοι αυτοί μέχρι σήμερα δεν έχουν επιτευχθεί πλήρω. Σήμερα ο πληθυσμό στην Ευρωζώνη γύρω στο 1% είναι πραγματικότητα και πολύ μακριά από τον στόχο που είχαμε θέσει αρχικά ως επιθυμητό και εσεί και ο πρώην πρόεδρο Ντράγκη, και ο πρώην Ντράγκη επανειλημμένως επαναλάβατε ότι η ε, ανάκαμψη τη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα εξαρτηθεί και από το κατά πόσον τα κράτη-μέλη εφαρμόσουν τι σωστέ δημοσιονομικέ πολιτικέ για να δώσουν κίνητρα για επενδύσει. Ωστόσο, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τα κράτη-μέλη που έχουν το περιθώριο για να κάνουν τέτοιες χρήσιμε διευκολυντικέ επενδύσει δεν το κάνουν γιατί ε, θέλουν απλώ να μειώσουν το δικό του εμπορικό πλεόνασμα. Αυτό που μας λείπει είναι ότι στην παράδο των ετών, μέσα στα χρόνια, έχει μειωθεί το ποσοστό των δημόσιων επενδύσεων. Και αυτό ιδίω στις χώρες όπου η ανάπτυξη είναι χαμηλότερη. Εκεί όπου οι επενδύσεις είναι μάλιστα ε, απαρχιωμένες. Ένας από τους βασικούς λόγους των χωρών αυτών να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς, να αντέξουν ε, στις κλιματικές αλλαγές, τα ε, δυσμενή καιρικά φαινόμενα. Εδώ λοιπόν υπάρχει η κατάρρευση, ή τουλάχιστον η συμπίεση της εσωτερικής ζήτησης και αυτό εμποδίζει την ανάπτυξη. Πιστεύετε λοιπόν ότι πέραν των εργαλείων που διαθέτει σήμερα η ΕΚΤ, μήπως χρειάζεται και νέα ε, νέα εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να σπρώξουν σε ανώτερα επίπεδα την ζήτηση στην Ευρώπη. Και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ποια θα ήταν αυτά τα νέα εργαλεία. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρατήρησή σας, για την πρώτη σας παρατήρηση. Απέχουμε πολύ ε, από τον σωστό στόχο του πληθωρισμού. Όμως πραγματικά είναι ένα θέμα συναρπαστικό εάν το σκεφτεί κανείς. Οι οικονομολόγοι πασχίζουν να το καταλάβουν ε, και το μελετούν. Σε πολλά μέρη του κόσμου ο πληθωρισμός ήταν χαμηλότερος από ό,τι αναμενόταν. Και πολλοί οικονομολόγοι και ειδικοί επιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει με την απομηχανή του πληθωρισμού. Ε, είναι ενδιαφέρον να παρατηρεί κανεί ότι ενώ έχει μειωθεί η ανεργία, η συμμετοχή στην απασχόληση έχει αυξηθεί, οι μισθοί όπως τους μετρούμε τέλο πάντων έχουν αυξηθεί και αυτοί, ωστόσο κανονικά θα έπρεπε να αυξηθούν και οι τιμές. περισσότερη ζήτηση που θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. Αλλά δεν συμβαίνει. Αυτό λοιπόν που μάλλον έχει γίνει και αυτό λένε οι εκλογικές επιφέρειες και αν παρατηρήσει κανείς ότι συμβαίνει στη χώρα του ή αλλού στην Ευρωζώνη, φαίνεται ότι οι εργοδότες αντί να αυξήσουν τις τιμές όπως τα έκαναν ε, χαρακτηριστικά, ουσιαστικά πιέζουν το περιθώριο. Ε, γιατί το κάνουν αυτό. Δύσκολο να το κατανοήσει κανείς ή να το αποτιμήσει. Επειδή αισθάνονταν ασφάλεια και βεβαιότητα, επειδή θέλουν να, να προστατεύσουν το μερίδιο της αγοράς τους κατά των ανταγωνιστών, επειδή δεν έχουν αρκετή εμπιστοσύνη στο πώς μπορούν να αντισταθούν ε, σε, άλλους, σε άλλες πηγές ανταγωνισμού. Δύσκολο να το πει κανεί. Αλλά αυτό παρατηρούμε προς στι στις αγορές. Τώρα θα διαρκέσει αυτό. Μεγάλο ερώτημα. Εάν οι παράγοντες αβεβαιότητας ε, πρετανεύσουν, εάν το Brexit ε, γίνει με τρόπο ομαλό, εάν η περίοδος μετάβασης είναι κατανοητή και εύληπτη, εάν η όλη η συζήτηση για τις αντίξωες συνθήκες στο εμπόριο οδηγήσει σε άλλο είδους διευθετήσεις με τους Κινέζους και τους Αμερικανούς. Εάν οι αριθμοί στην Κίνα τα πάνε πάλι καλύτερα. Είναι πολλά τα στοιχεία από μακροοικονομικής σκοπιάς που πρέπει να τα δούμε, αλλά εάν αυτά συμπέσουν, τότε μπορεί να οδηγήσουν τους οργοδότες να διοχετεύσουν στις τιμές την αύξηση του κόστους που αντιμετωπίζουν. Αυτό θα είναι κρίσιμο για τον αριθμό και τα στοιχεία του πληθωρισμού, όμως προς στιγμή αυτά παρατηρούμε. Τώρα για τις υπόλοιπες πολιτικές είπα όσα είχα να πω για το δημοσιονομικό μέτωπο. Η νομισματική πολιτική ε, μεταφέρεται και εφαρμόζεται καλύτερα όταν και άλλοι πολιτικοί φύνοντες αναλαμβάνουν το δικό τους μερίδιο. Σε κάποιες χώρες με δημοσιονομικό περιθώριο παρατηρείται ότι σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν αυτό το περιθώριο για καλούς σκοπούς ιδίω σε ένα μέλο τη Ευρωζώνη που μου έρχεται στο νου. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι ευπρόσδεκτο από εμά. Σα ευχαριστούμε ο κύριο Γιουτζίκα, του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να τηρήσω τους κανόνες που έθεσε η Πρόεδρός μας, οπότε θα Έχω μία ερώτηση προς την κυρία Λαγκάρτ. Όσον αφορά τη δημοσίευση αναλύσεων για τις παρενέργειες της τρέχουσας ε, νομισματικής πολιτικής. Αυτό θα σας το ρωτήσω την επόμενη φορά. Τώρα θα σας ρωτήσω για το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στο ΕΚΤ και του σώματος των εποπτών. Ο κύριος Ντράγκη στην Επιτροπή μας την προηγούμενη φορά απάντησε λέγοντας ότι το στοιχείο κλειδί ήταν κατά πόσο θα μπορούσε να κρυθεί όχι μόνο η ρύθμιση και η διαχείριση, αλλά και η αποτελεσματικότητα του έργου της ΕΚΤ. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών πιστεύετε ότι τώρα ασχολείται με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΚΤ ή όχι. Σας ευχαριστώ. Το ελεκτικό συνέδριο, συγγνώμη, το ελεκτικό συνέδριο. Ναι, ναι, όσον αφορά ε, την ε, διαχείριση της ΕΚΤ είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, η αποτελεσματικότητα όντως ελέγχεται ανεξάρτητα από το ελεγκτικό συνέδριο όπως προβλέπεται από τις συνθήκες. Αυτό όσον αφορά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Τώρα το έργο του Ελεκτικού συνεδρίου είναι ένα έργο το οποίο εγώ θα στηρίξω να ξέρετε. Θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που χρειάζονται για να επιτελέσουν το έργο τους, αλλά συγχρόνως οι αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τη, αυτό που ονομάζετε εσείς φαντάζομαι πολιτικές ε, της ΕΚΤ, αυτό είναι ένας ρόλος της ίδιας της ΕΚΤ και που είναι κάτι διακριτό και διεξάγεται με απόλυτη ανεξαρτησία έτσι όπως προβλέπεται και από το καταστατικό της ΕΚΤ. Ευχαριστώ πολύ. Καρολάιν Νάτιγκαλ, Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαγκάρτ. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια για τον ορισμό σας. Θα συνεχίσω στα Ολλανδικά. Μπορεί να μην είναι τόσο ευχάριστο, αλλά ναι. Λοιπόν, ζούμε ενδιαφέροντες καιρούς με πολλές προκλήσεις και είναι πολύ σημαντικό το δικό σας έργο, είναι και μια πρόκληση σταθερότητα τιμών. Πρέπει να φροντίσουμε επίσης για την ευημερία του ευρώ. Υπάρχει ανεξαρτησία της ΕΚΤ που είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να παραμείνει. Όμως ανησυχώ λίγο για τις διάφορες πολιτικές της ε, ΕΚΤ. Ήδη και την προηγούμενη φορά είδαμε ότι μειώθηκαν τα επιτόκια, που σημαίνει ότι οι καταθέτες, οι αποταμιευτές δεν κερδίζουν τίποτα από τις αποταμιεύσεις τους, για να μην πω ότι πρέπει να πληρώσουν και από πάνω. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, έχουμε μεγάλα ταξιδιωτικά ταμεία, πολύ σημαντικά, αλλά εδώ με τα χαμηλά επιτόκια ρωτάω γιατί επιμένει η ΕΚΤ στο στόχο του 2% και δεν θα έπρεπε να μείνει ανοιχτή να δει το θέμα της σταθερότητας μόνο και αλλιώς. Τα τελευταία 16 χρόνια πράγματι έχουν συμβεί πάρα πολλά και στην Ολλανδία υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την πολιτική της ΕΚΤ γιατί τα συνταξιδοτικά ταμεία θα πρέπει να ευημερούν και αυτά. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για όλα αυτά. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η ΕΚΤ δεν ξεχνάει τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπο των πολιτικών της. Είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε, τις επιπτώσεις δηλαδή των πολιτικών μας. Τώρα, Δεν μπορεί να τέθεται το ζήτημα η μία κατηγορία ή η άλλη κατηγορία. Πρέπει να ασχοληθούμε γενικότερα με τον αντίκτυπο της πολιτικής μας για τη στήριξη της ανάπτυξης, για την ενθάρρυνση των επενδύσεων, για να επωφεληθούμε από το χαμηλό κάστος χρηματοδότησης, να ασχοληθούμε με την απασχόληση ε, στην Ευρωζώνη. Η ΕΚΤΕ προσπαθεί να τηρήσει την εντολή της και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της οικονομίας. Οπότε αυτά είναι που μπορεί να κάνει. Φυσικά και υπάρχουν παρενέργειες και πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας και πρέπει και να τις προλαβαίνουμε αν γίνεται. Το σύστημα των δύο βαθμίδων που καθιδρύθηκε το Σεπτέμβριο είχε ακριβώς αυτό το στόχο να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να προσφέρουν μηδενικό επιτόκιο αντί για αρνητικό και άρα να συνεχίζουν έτσι να χρηματοδοτούν την οικονομία. Ε, ξέρω ότι για ορισμένα ταξιδιωτικά ταμεία σε κάποιες χώρες αυτό είναι πρόβλημα και θα είμαστε πολύ προσεκτικοί γι' αυτό και θα δούμε πόσο καλύτερα μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας αυτούς τους παράγοντες στην αναθεώρηση της στρατηγικής μας. Ευχαριστούμε. Πιέρ Νικολά Πεντατσίνη, μία γεγραμμένος παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα τα πω Ιταλικά. Ευχαριστώ. Ε, Πρόεδρε Λαγκάρντ. με τις αλλαγές τελευταίας στιγμής, τις μετατάξεις τελευταίας στιγμής, το επόμενο Συμβούλιο 13 Δεκεμβρίου και ε, για τους αρχηγούς κατών και κυβερνήσεων που έχουν συμφωνήσει τον ε, μηχανισμό σταθερότητας, θα πρέπει να ξανασυζητήσουν την ε, δική σας, το δικό σας εσωτερικό καταστατικό. Χώρε όμως όπως η Ελλάδα δεν διασώθησαν όπως μας έδειξε το παρελθόν, αλλά κυρίως η Τράπεζα της Γαλλία και τη Γερμανίας ήταν εκτεθειμένες ε, στην ε, Ισπανία και Ελλάδα. Και χώρε όπω η Ιταλία βρέθηκαν εκτεθειμένε με 10 δι που δεν επέστρεψαν ποτέ. Εδώ λοιπόν, σε περίπτωση τραπεζική κρίση, υποτίθεται ότι με την Τραπεζική Ένωση δεν υπάρχει παρέμβαση, αλλά προτείνεται και δημοσιονομική γραμμή ενισχυμένη που θα διευκολύνει τα κράτη με δημόσιο χρέος το οποίο θα θεωρείται μη βιώσιμο. Παράδοξο αυτό, αλλά μπορεί να γίνει αποδεκτό. Οι τράπεζες που αντιμετωπίζουν κρίση όπως η Deutsche Bank και οι χώρες όπως η Γερμανία που δεν έχουν ανάγκη ε, θα έχουν πρόσβαση, ενώ οι χώρες που έχουν ανάγκη δεν θα έχουν πρόσβαση και θα πρέπει να συνεισφέρουν για να καλύπτουν τα κεφάλαια και τις απώλειες των άλλων. Ποια είναι λοιπόν η άποψή σα για αυτό το μηχανισμό ε, τη ε, σταθεροποίηση ω συστημικού εργαλείου για να αντιμετωπίζονται οι κρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Θα είμαι εντελώς ξεκάθαρη για τον ESM, για το μηχανισμό σταθερότητας. Γιατί νομίζω ότι εδώ γνωρίζω και ξέρω γιατί μιλάω. Ήμουν ε, και στην αίθουσα όταν λήφθη η απόφαση για τη δημιουργία του. Η λειτουργία του ΕΣΜΑ αυτή τη στιγμή σκοπό έχει να ενισχύσει το σύστημα διαχείρισης κινδύνου της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει κανένα θέμα για μένα Τέτοιου είδου προτάσει θα υποβληθούν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αργότερα μέσα στο μήνα. Και ξέρω ότι αυτό προκαλεί έντονε συζητήσει σε πολλέ χώρε, όμω ο σκοπό είναι ακριβώ να αντιμετωπίσει το θέμα της ευπάθειας της ευπάθειας και του ε, οικονομικού κινδύνου. Γι' αυτό πρέπει να ανασυγκροτηθεί ο ΕΣΜ και να ε, ενισχυθεί όπως ήδη συζητιέται. Όμως ε, τα εργαλεία συλλογική δράση που κάποιους τους έχουν ε, συνταράξει, είναι κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε κάνει ό,τι μπορούσε για τα, είχε, είχε κάνει μπορούσε για τα εργαλεία κοινή δράσης, συλλογική δράσης. Είναι εργαλεία έκδοση που έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι αν υπάρξει στόχευση, οι μέτοχοι με τις λιγότερες μετοχές δεν μπορούν να κρατούν όμοιρο στους υπόλοιπους μετόχους για τα δικά τους ίδια συμφέροντα. Είναι δηλαδή ένας τρόπος να προστατεύεται η πλειονότητα στις ε, ατασταλίες μιας μειοψηφίας. Αυτό δεν έχει να κάνει αναγκαστικά με την Ευρωζώνη, είναι μια ε, διάταξη που θα ισχύει παγκοσμίω εφόσον υπάρχουν τέτοιου είδου ελλείψει ισορροπία. Για να μπορούμε να διαχειριστούμε κρίσει. Όχι για να πάρουμε κανενό τα υπάρχοντα, ούτε να φανούμε εχθρικοί προ κάποια, εχθρική προς κάποια χώρα, το ανάποδο. Η κυρία Μάρκες από το Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σήμερα η συζήτηση για τις κλιματικές αλλαγές φλένεται να είναι ε, το βασικό θέμα και μόλις ξεκίνησε η COP στην Μαδρίτη. Ε, στην προηγούμενη ακρόασή σας στο Ευρωκοινοβούλιο, εδώ σε αυτή την αίθουσα, ανακοινώσατε ότι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών θα γίνει παντιέρα σας, θα γίνει από τις προτεραιότητες της ΕΚΤ. Οι κλιματικές αλλαγές έχουν επίσης κοινωνικές και μακροοικονομικές συνέπειες, όπως μόλις ε, ακούσαμε. Οι κλιματικοί κινδύνοι έχουν εντοπιστεί από την ΕΚΤ ως ένας από τους βασικούς κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν το τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης και την ε, λειτουργία της οικονομίας του. Ε, την ε, εντολή τη, η ΕΚΤ έχει κάθε νομιμοποιήσει, κυρία Λαγκάρτ, για να υποστηρίξει ενεργώ τη μετάβαση σε μια ουδέτερη ε, από πλευρά άνθρακα οικονομία. Μπορεί να βοηθήσει να οριστούν οι σωστοί κανόνε και να εφαρμοστούν. Από εμά θα έχετε όλη την απαραίτητη στήριξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι περιβαλλοντικέ προτεραιότητε είναι το βασικό τμήμα των προτεραιοτήτων τη και του προγράμματο εργασία τη. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για τι κατεπίξουσε ανάγκε των κλιματικών αλλαγών και θα τα συζητήσουμε και στην επόμενη Ολομέλεια. Η αναθεώρηση της ε, Νομισματική πολιτικής στρατηγικής δεν μπορεί να παραβλέψει αυτή τη διάσταση. Ερωτήσεις. Θα ε, ε, αντιμετωπίσετε σίγουρα φραγμού. Η ερώτησή μου είναι πώς θα υπαρπηδήσετε αυτά τα εμπόδια, πώς θα πείστε του συναδέλφου σας των άλλων κεντρικών τραπεζών που θεωρούν ότι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών ε, είναι θέμα της δημοσιονομικής πολιτικής και όχι της νομισματικής. Και τι συγκεκριμένα μέτρα σκέφτεστε να προτείνετε για να υλοποιηθούν ως προς τις ε, εσωτερικές συναλλαγές και ενέργειες της ΕΚΤ, αλλά και διεθνώς στις σχέσεις της ΕΚΤ. Εδώ εννοώ ότι συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να υπολείστε στο G7, στο G20, στις σχέσεις με την Κίνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι συνοπτικότατη στην απάντησή μου, διότι πραγματικά νομίζω ότι ήδη το έχω απαντήσει. Πρώτα απ' όλα από τη σκοπιά της ανάλυσης και μετά από τη σκοπιά της εποπτείας και τη σχετική μα αρμοδιότητα. Και τρίτον, με τι άμεσε επενδύσει και τη διαχείριση των συνταξιδοτικών ταμείων. Τέταρτον, με τα προγράμματα βάσει των οποίων λειτουργούμε ε, και τα οποία χειριζόμαστε και πρέπει να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε πόσο κλιματικέ αλλαγέ μπορεί να έχουν κάποιο αντίκτυπο στι αξιολογήσει κινδύνου που εκδίδουμε. Εδώ πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε δραστήριοι σε πολλά φόρουμ ταυτόχρονα. Είμαστε μέλο του δικτύου των κεντρικών τραπεζών και των εποπτών για, την, για το πρασίνισμα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Όπως ξέρετε, στη φάση αυτή εδώ ε, ε συνεργάζονται τουλάχιστον 50 κεντρικέ τραπεζέ με του διευθυντέ του και τους συνεργάτες τους Οπότε κινούμαστε ε, σαφώς προς τις ε, ενέργειες πρασινίσματος. Είμαστε εξίσου ενεργοί στο G7 με τον Μπενουά Κερέ που πρόσφατα εξέδωσε μια σχετική έκθεση με τέτοιες θετικές ε, προς την κατεύθυνση που αναφέρετε και εσείς απόψεις. Κάθε φόρουμ στο οποίο ε, υπάρχουμε και έχουμε παρουσία, το G20 είναι επίσης ένα από αυτά όπου θα συζητηθούν οι κλιματικές αλλαγές, οπωσδήποτε. Και εκεί ε, κοιτάζουμε να σωματώσουμε όλες αυτές τις παραμέτρους. νομίζω ότι είναι πολύ... Ο Μπενουά είναι πολύ ε, ένθερμος για την αντιμετώπιση των κλιματικών ελλαγών. Πολύ περισσότερο από ό,τι έχει φανεί εδώ, αλλά και στο G7 και στο G20 θα γίνει ό,τι ε, πρέπει. πάντω να είστε βέβαιοι ότι είναι υπέρ, υπέρμαχος της καταπολέμησης των κλιματικών ελλαγών. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα-δύο λεπτά ακόμη για ένα τελευταίο Catch the Eye. Have... Θα είναι ο κύριο Καστάλντο, μη Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, τη Λακάρτ. Είναι διχασμένο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤΑ για τη μελλοντική νομισματική πολιτική. Υπάρχει θέμα αξιοπιστίας και θέμα δυνατότητας επιρροής. Οι επενδυτές θέλουν κάποιο μήνυμα από την ΕΚΤ. Ένα από τα επιτεύγματα του κυρίου Ντράγκη μέχρι πρόσφατα ήταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μιλούν με μία φωνή υπήρχε συνένεση και ήταν αυτό ζωτικό σημείο. Ήδη όταν ο κύριος Ντράγκη είπε ότι θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, καταφέραμε όντως και αποφύγαμε ε, παρετέρω κρίση. Και ακριβώς λοιπόν χρειάζεται στήριξη της οικονομίας στο μέλλον και χρειάζεται και πειθό προς τις αγορές και τους επενδυτές πρέπει να μην δίνουμε την εντύπωση ότι έχει περιορισμένα περιθώρια ελιγμών η ΕΚΤ, γιατί αλλιώς τότε το βάρος της νομισματικής πολιτικής θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Στη νομισματική πολιτική μάλλον. Οπότε ρωτάω, είναι διχασμένο το Δικαιωτικό Συμβούλιο και τι σημαίνει αυτό για το μέλλον. Θα κάνετε τη ζωή μας πιο δύσκολη και τι θα κάνετε ώστε να γιατρευτούν αυτές οι πληγές και να είναι ενιαία η φωνή του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν θα σας εκπλήσει η απάντηση να ξέρετε ότι υπήρξε ομόφωνα συμφωνία για τη συνολική εντολή και τους στόχους μας. Όλα τα μέλη λοιπόν ομόφωνα δεσμεύονται να πετύχουν τον στόχο της σταθερότητας τιμών. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης ήταν ομόφωνο για την ανάγκη να προσθεθούν και άλλες νομισματικές διευκολύνσεις. Οι διαφορές είχαν να κάνουν με τη στάθμιση, την ακριβή στάθμιση και με το είδος των μέσων που θα χρησιμοποιούσαμε. Αλλά αυτή είναι μια πολύ τεγή συζήτηση και σίγουρα οδηγεί μπροστά και συνάδει με τις δικές μου ιδέες για διακυβέρνηση. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ εννοείται για να επιτευχθεί συνένεση για το πακέτο όταν καταλήξουμε και χρειαστεί ένα τέτοιο πακέτο. Αν υπάρξουν διαφωνίες, θα υπάρξουν διαφωνίες. Και θα πρέπει να βρούμε ένα υγιή και αποτελεσματικό τρόπο να το χειριστούμε. Υπάρχουν πολλές κεντρικές τράπεζες που χειρίζονται τέτοια ζητήματα. Ωραία, είναι ιδανικό το να υπάρχει ευρεία συνένεση. Αλλά η έκτη είναι αρκετά ισχυρή και τη φήμη της την έχει κερδίσει ακριβώς γιατί μπορεί να αντέξει και διαφωνίες άπαξ και αυτές υπάρχουν. Σας ευχαριστώ θερμά. Έτσι ολοκληρώνεται ο νομισματικός μας διάλογος. Ε, ευχαριστώ όλους τους ευρωβουλευτές που συμμετείχαν. Σας ευχαριστώ κυρία Λαγκάρτ. Δεδομένου ότι ήταν ε, ο πρώτος διάλογος ε, μετά από τέσσερις μόλις εβδομάδες, είχαμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε και θα έχουμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αφήνω την Προεδρία στον κύριο Νίτερμαγερ. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ καθίστε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε ακόμη κάποια θέματα στην ημερήσια διάταξη. Προχωράμε στο σημείο 5. Οι οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η έκθεση 2019. Ο εισηγητής μας είναι ο Μπάς Έικχαουτ από τους Πρασίνους. Χωρίς πολλά πολλά, λοιπόν, θα σας δίνω πέντε λεπτά για να μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ίσως να μην χρειαστώ και τα πέντε λεπτά. Είναι η πρώτη δήλωση της Επιτροπής ΕΚΟΝ για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, η επί της αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ε, εμείς γνωμοδοτούμε. Γι' αυτό είναι σύντομο το κείμενο. Έχουμε περιορισμό όσον αφορά τον αριθμό ε, γραμμάτων, τον αριθμό ψηφίων μιας ε, τυπογραφικών χαρακτήρων και είναι σύντομη για το λόγο αυτό, αλλά με γνωμοδοτήσεις μπορούμε να πούμε κάποια θέματα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία σίγουρα θα πρέπει να θίξουμε. Τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, στην αύξηση των επιπέδων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι το επίπεδο επενδύσεων είναι πιο χαμηλό από ό,τι πριν την κρίση λοιπόν ε, σημαντικό να αυξηθούν οι επενδύσεις αυτές. Πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι υπάρχουν αλλαγές που συνεχίζονται στην ΕΤΕ. Πολύ θα θέλαμε να γίνει μια κλιματική τράπεζα η ΕΤΕ. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά βέβαια πρέπει να μεταφερθούν και να γίνουν ε, πραγματική δράση και αν μη τι άλλο να έχει η ΕΤΕ μια σωστή μεθοδολογία ώστε να συμπεριλαμβάνει στους στόχους της το να υπάρξει πιο ξεκάθαρα διατυπωμένη ευθυγράμμιση με τους κλιματικούς στόχους για να γίνει μια κλιματική τράπεζα. Υπάρχει επίσης το σχέδιο Juncker. Και φυσικά και πρέπει να συζητήσουμε για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ σημαντικός ο στόχος του να καταλήξουμε σε υψηλό ποσό. Αλλά βέβαια το χάσμα των επενδύσεων πρέπει να κλείσει και πρέπει να ξέρουμε τι στόχους θέλουμε να πετύχουμε. Μερικές φορές μπορεί να πρέπει να υπάρξει και ένα παζάρεμα και μπορούμε να το συζητήσουμε. Σίγουρα γιατί η ΕΤΕ στις μελλοντικέ επενδύσεις και στο επόμενο σχέδιο που θα μας έρθει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο που θα ονομάζεται ε, σχέδιο βιωσιμότητας. Τέλος, λέμε στη γνωμοδότηση για την διαφάνεια. Και αυτό έχει να κάνει και με τις συζητήσεις που λένε πώς θα είμαστε σίγουροι για την προσθετικότητα Πρόκειται για μια δημόσια τράπεζα επενδύσεων η ΕΤΕ και υπάρχουν πάρα πολλέ επενδύσεις που συνεχίζονται. Πώς λοιπόν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει προσθετικότητα. Να μην είναι απλώς μια παραπάνω ιδιωτική τράπεζα, αλλά να έχουμε μια δημόσια τράπεζα και άλλα πράγματα θα μπορούσαμε να βάλουμε στη γνωμοδότηση και ευχαρίστω να τα προσθέσω. Αλλά τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να περιορίσουμε το μέγεθο τη γνωμοδότηση. Αλλά με τι τροπολογίε θα μπορέσουμε να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία. Συμφωνούν πάντω και οι σκιώδει και πρόκειται για γνωμοδότηση προ την Επιτροπή Προπολογισμών. Και θα ήθελα να ακούσω αντιδράσει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και από του άλλου συναδέρφου εννοείται. Και να καταλήξω σε μια γνωμοδότηση με ευρεία συνένεση, ώστε η γνωμοδότησή μας να ληφθεί υπόψη από την ε, Επιτροπή Προπολογισμών. Ευχαριστούμε, Μπά. Ε, τώρα έχουμε του σκιώδει εισηγητέ. Πρώτα από το ΕΛΚΑ, ε, η κυρία Φιτσέρελ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει πάνω στο θέμα αυτό. Ε, αναφέρεται σε κάποια από τα βασικά θέματα στα οποία έχει επικεντρωθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, το τελευταίο έτος ε, και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια από αυτά. Επικροτώ το ότι ε, θέλει, πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει επαρκή κεφαλαιοποίηση τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ότι θα πρέπει να συνάδει με του στόχου τη Συμφωνία του Παρισίου πριν το τέλο του 2020, καθώ και το ότι επικεντρώνεται στη διαφάνεια. Το σχέδιο γνωμοδότηση επικεντρώνεται στην κλιματική χρηματοδότηση και νομίζω ότι αυτό ενδείκνυται δεδομένη τις κρίσεις που αντιμετωπίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει μακρά ιστορία όσον αφορά τη χρηματοδότηση τη κλιματική δράση. Πριν 10 χρόνια έπαιξε ρόλο πρωτοπόρου ε, με το πρώτο ομόλογο κλιματική ε, συνείδηση. Επίσης ε, αναφέρεται η προσήλωση της κυρίας Φοντερ Λάιεν, η ε, τράπεζα Επενδύσεων ε, να γίνει κλιματική τράπεζα. Αυτό είναι σημαντικό στόχο για να πετύχουμε τους ε, στόχους μας όσον αφορά το κλίμα. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πτυχές που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, όπως είναι η προώθηση της επένδυσης στην Ευρώπη, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η υποστήριξη της ψηφιακής οικονομίας. Και αυτοί είναι όλοι οι τομείς που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ως Επιτροπή. Ε, η έκθεση για το 2019 τονίζει το γεγονός ότι οι επενδύσεις ε, στην, ε, στις υποδομές βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα τα τελευταία 15 χρόνια και ότι επίσης χρειάζονται περισσότεροι πόροι για την ψηφιακή μετάβαση. Από την οικονομική κρίση και μετά είχαμε σίγουρα μια δεκαετία ασθενούς επένδυσης και θα πρέπει να ε, ε, λάβουμε υπόψη μας τις βασικές υποδομές όπως είναι η στέγαση θα πρέπει να συνεχίσουν να παραμένουν αυτοί οι βασικοί στόχοι τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη γνωμοδότηση με κάποιο τρόπο. Θα πρέπει επίση ε, να ε, ε, σημειώσουμε πόσο σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τι κλιματικέ τη επενδύσει να τι συνοδεύσει από μέτρα δικαιοσύνη ώστε να μην μείνει κανεί πίσω. Επίσης, όσον αφορά τον κοινωνικό αντίκτυπο. Ε, δεν θα πρέπει να ε, ε, έχουμε δείκτες μόνο οικονομικούς όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ιδιαίτερα διότι θέλουμε να αυξήσουμε τι επενδύσει στην Ευρώπη και να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάντως θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ καλή γνωμοδότηση αυτή ε, και συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τον ε, εισηγητή. Ευχαριστώ, Γιώχημ Σούστερ. Θα μιλήσω γερμανικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι αναφέρονται πολύ σημαντικά θέματα στη γνωμοδότηση, τα οποία συμμεριζόμαστε. Τρία-τέσσερα σημεία θα ήθελα να τονίσω εδώ, τα οποία είναι σημαντικά για μας. Ε, καταρχάς, αυτό που είπε ήδη ο εισηγητής, ε, επικροτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διευρύνει τις επενδυτικές της δραστηριότητες ε, ώστε να καταστεί κλιματική τράπεζα. Το θέμα είναι βέβαια αυτό στην πράξη τι σημαίνει ακριβώς, σε ποιες επενδύσεις θα μπορούν να προωθηθούν και ποιες όχι. Και με τι ε, εργαλεία θα μπορέσουμε να ε, στηρίξουμε τις επενδύσεις αυτές. Το άλλο θέμα είναι ότι δεν μας ενδιαφέρουν εδώ μόνο οι ιδιωτικές επενδύσεις, μας ενδιαφέρουν και οι δημόσιες επενδύσεις, ιδιαίτερα από δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις. Διότι το ότι έχουμε τέτοια έλλειψη επενδύσεων οφείλεται και ε, στις κρατικές επενδύσεις και τον συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, ε, τις επενδύσεις αυτές ε, θα πρέπει να τις αφαιρούμε από το χρέος, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ε, όσον αφορά την κοινωνική διάσταση και τα σχετικά προγράμματα, επειδή θέλουμε να προωθήσουμε μια οικολογική μετάβαση, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τον κοινωνικό αντίκτυπο αυτών. Επίσης, θα πρέπει η περιφερειακή κατανομή να γίνεται και σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια. Το τέταρτο θέμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας είναι ότι χρειαζόμαστε αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει περισσότερο λέγιν και τα συμπεράσματα του ελεγκτικού συνεδρίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων ε, θα πρέπει να ληφθούν επίση υπόψη στην δομή διακυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πάντω, ε, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε πολύ επικοδομητική συζήτηση και Ελπίζω έτσι να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε ώστε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κινηθεί προς την σωστή κατεύθυνση στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ ε, από το ΡΙΝΙΟΥ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Έικχαουτ και τους συνεργάτες του για την καλή δουλειά που έχουν κάνει πάνω στη γνωμοδότηση αυτή. Θα ήθελα να επισημάνω κάποια ε, σημασία θέματα, τα οποία όμως θα ήθελα να συμπεριληφθούν στην γνωμοδότηση αυτή. Νομίζω ότι και οι συνάδελφοι εδώ θα συμφωνήσουν μαζί μου. Θα ήθελα καταρχάς να δράξω την ευκαιρία για να τονίσω τη σημασία της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με άλλους εταίρους. Αυτό τονίστηκε στο επιχειρησιακό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως το 2019. Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη συνεκτικότητα στη συζήτηση αυτή, δεδομένου ότι θα έχουμε μια σειρά παραγόντων ε, στο μέλλον που θα συμμετέχουν ε, στις εργασίες. Δεύτερον, η γνωμοδότηση αναφέρεται ε, στην μετατροπή της Τράπεζα Επενδύσεων σε Κλιματική Τράπεζα και τους στόχους του Παρισιού. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε και το μελλοντικό Green Deal, την Πράσινη Συμφωνία. λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και το πώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήδη έχει αρχίσει ε, την μεταρρύθμιση. Επίσης, όσον αφορά το InvestEU, ε, όπως ε, αναφέρθηκε. Υπάρχουν επενδύσεις ε, που εμπίπτουν στην κατηγορία των κοινωνικών επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Θα θέλαμε όμως εδώ να συνδέσουμε περισσότερα τα θέματα αυτά, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τον αντίκτυπο των επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήδη στο πλαίσιο του ΕΦΣΥ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, εφαρμόζει τέτοιου είδους επενδύσεις. Είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό κατά νου. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό είναι ότι τοπικοί φορείς σε, διάφορα μέρη της Ευρώπης ε, έθιξαν το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό να υπάρχουν γραφεία συνδέσμου ε, για να ενισχυθεί η συνεργασία με ιδιώτες και δημόσιους φορείς με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και να τους ενημερώνει σχετικά με το φάσμα οικονομικών δυνατοτήτων, δυνατοτήτων επένδυσης που έχουν στη διάθεσή τους. Νομίζω ότι αυτό θα μπορέσει να βελτιώσει την γνωμοδότηση. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να αυξήσει τις δραστηριότητές της σε τοπικό επίπεδο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ θερμά για τη δυνατότητα συνεργασίας που έχουμε και προσβλέπω στην καλή συνεργασία με τον κύριο Έικχουτ και την ομάδα του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. ID δεν έχει. ECR. Παρακαλώ, κυρία Καστικνόν. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για την καλή αυτή, το σχέδιο γνωμοδότηση. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει τεράστιες δυνατότητες, αλλά διαφέρουμε και σε κάποια σημεία. Η γνωμοδότηση λέει ότι θα έπρεπε να γίνει κλιματική τράπεζα η ΕΤΕ. Αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι αυτό σημαίνει πολιτικοποίηση παρετέρω της ΕΤΕΠ. Για τη βάση πολιτικής ατζέντα θα προωθούνται οι πόροι και όχι για την ανάπτυξη και την απασχόληση παντού στην Ευρώπη. Εάν λοιπόν παρέκλεινα από το στόχο της η ΕΤΕΠ υπέρ του κλίματος, αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτά για διαφορετικούς σκοπούς στο μέλλον. Κάτι το οποίο ανοίγει το κουτί της Πανδώρας. Η επενδύσεις που πηγαίνουν τώρα σε στερεά καύσιμα που θα έπρεπε να σταματήσουν σύντομα. Εδώ θέλω να ρωτήσω πρώτον, αυτό το εμπάργο επενδύσεων θα αφορά και την συντήρηση ή θα αφορά μόνο την επέκταση σε νέα προγράμματα. Δεύτερον, όπως όλοι γνωρίζουμε υπάρχουν πολλές περιοχές στην Ευρώπη που εξαρτώνται από την παραγωγή ορυκτών ε, καυσίμων και χρειάζονται βοήθεια στην μετάβαση. Θα υπάρχουν αρκετές πράσινες επενδύσεις μέχρι τα τέλη του 2020 στις περιοχές αυτές για να αντικαταστήσουν τα ορυκτά. Επίσης θέλω να επενθυμίσω σε όλους ότι υπάρχουν διάφορα σκοτεινά σύννεφα στον ορίζοντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει έναν από τους βασικότερους εισφορείς της ήδη από τον επόμενο μήνα. Ευχαριστούμε τέλος από την ΓΚΟΕ. Έχουμε την κυρία Μπρή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για την σύνταξη αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης. Πάει στη σωστή κατεύθυνση, βάζοντα το δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης στην ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τώρα σχόλιο ένα εδάφιο για την πρώτη παράγραφο. Η έκθεση θα πρέπει να ακολουθεί ε, συνεπέστερη προσέγγιση για τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οικολογική μετάβαση. Η τελευταία έκθεση της δημοσιονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφιστά την προσοχή ε, στο 3% ε, που δεν έχει επιτρέψει όμως παρόλα αυτά να ξεκαθαριστούν καλύτερα τα κρατικά δημοσιονομικά. Θα πρέπει λοιπόν ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνεισφέρει στην αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η έκθεση τονίζει προβολικά τα δημοσιονομικά κριτήρια. Στι 2 και 3 Προφανώς συμμεριζόμαστε την δική σας την άποψη για την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αφιερώσει ένα κομμάτι των κονδυλίων τη στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, αλλά χρειάζονται κάποιε διευκρινήσει. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα προβλέπεται στο 2021. Αυτό πρέπει να το χαιρετήσουμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε και σε επιφυλακή Δεύτερον, σε, από την πλευρά της συνέπειας θα πρέπει να δούμε εάν η ΕΤΕ μπορεί να ορίσει και οικολογικά κριτήρια για τα χαρτοφυλάκια των προϊόντων της. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κοιτάξουμε μήπως μπορούμε να επηρεάσουμε το κείμενο ακόμη και μπορούμε να βάλουμε την έγκρισή του μας το 2021 και για την παράγραφο 4 η ΕΤΕ δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στο κλίμα, αλλά να θέσει και στόχου κοινωνική δικαιοσύνη. Θα πρέπει να υπάρξει μια κοινωνικώ υπεύθυνη στάση για να απογορευτούν παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ω προ αυτό, προτείνουμε η ΕΤΕ να ενισχύσει το, ε, την αρμοδιότητα εποπτείας που έχει, κάνοντας εξάντια αξιολόγηση των κρατών για να εντοπίσει τα ε, τον κίνδυνο του κάθε προγράμματο όρφου στα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει επίση να ασχοληθεί και με την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Και εντό των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κατανέμοντα ε, σωστά τη χρηματοδότηση μεταξύ των διαφορών περιοχών, αλλά και ε, προωθώντα τι καινοτόμε οικολογικέ επιχειρήσει παρά του μεγάλου διεθνεί ομίλου. Ε, για την ε, φορολογική αδικία είδαμε με κυβερνητικές οργανώσεις να ε, μιλούν για την ανάγκη η να υποστηρίξει προγράμματα που θα προστατεύουν από την άνθηση των φορολογικών παραδείσων. Υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα που είχαν σχέση με, τον, με τη Μονσάτο Φορσέκα και το Panama Papers. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ε, δυνατότητες ε, χρήσης δικτών συγκριτική αξιολόγηση για να ε, αποφεύγουμε την αναδρομή σε φορολογικού παραδείσους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα κατάλογο, ένα αρνητικό κατάλογο φορολογικών παραδείσων από το τίποτα είναι καλύτερο ακόμη και αν έχουμε διασμούς. Θα πρέπει λοιπόν το 50% των φόρων να είναι λιγότερο αλλά όχι βάσει των κανόνων CFC ε, και να ολοκληρώσω το σχόλιο με τελευταία παράγραφο. Θέλουμε μια ΕΤΕ πιο διαφανή. Προφανώς ε, το σημείο αυτό ε, καλώς υπάρχει στην έκθεση. Πρέπει να υπάρξει και αναθεώρηση των κατερίων όμως για την καταπολέμηση της εξαπάτηση και της τη κατάχρηση και τη απάτη, μάλλον, και ότι τα κριτήρια των σκανδάλων διαφθοράς όπως της Volkswagen. Με τη χρήση λογισμικών σε καταστάσεις εργαστηρίου για να μπορεί η εταιρεία να ξεγελάει τα τεστ και να τα, υπερβέ, να τα υπερπηδήσει, ε, όλα αυτά δεν πρέπει να επιτραπούν ξανά. Πρέπει να αξιοποιήσουμε και τη λειτουργία του Όλαφ και του Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να βεβαιωθούμε ότι ε, οι ανθρώπινοι πόροι και απαραίτητοι δημοσιονομική πόροι αφιερώνονται στις ανακριτικές διαστηριότητες της ε, ΕΤΕ. Μάλιστα, σήμερα παίρνετε βραβείο μακροσκελέστατης ε, παρέμβασης. Στο Catch the Eye έχουν γραφεί ο κύριος Ρολά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ένα από τα θέματα που ζήτησα πρόσφατα με κάποιους από την ΕΤΕΠ είναι όταν προτείνεται μια κλιματική ατζέντα από πάνω προς τα κάτω υπάρχουν πολλά και να και είδαμε ήδη την αυτοκινητοβιομηχανία που ανακοίνωσε 40.000 απώλειες για τελικά ε, η εσωτερική καύση θα αντικατασταθεί από ηλεκτρικά οχήματα. πρόθεσμα το κόστος είναι μεγάλο και χρειάζεται χρηματοδότηση είτε από την ΕΤΕΠ είτε από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Οπότε ρωτάω τα δικά τους τα ομόλογα πόσο θα πάνε στην συνοχή. Ε, ρώτησα, δεν μου είπαν όμως και όταν πρόκειται επίσης και για δάνεια ή για αγορές ενεργητικού, για την δίκαια μετάβαση ή για την αντικατάσταση θέσεων απασχόλησης που χάνονται. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα καλύψουμε όλα αυτά. Οπότε η μεγάλη μου ανησυχία με την ΕΤΕΠ είναι ότι θα αυξηθούν τα δάνεια και για το Ηνωμένο Βασίλειο είμαστε εκτεθειμένοι με 36-37 δισεκατομμύρια για 12 χρόνια στην ΕΤΕΠ. Και αυτή είναι μεγάλη μου ανησυχία. Και πολύ θα ήθελα αυτό να αντιμετωπιστεί στις συζητήσεις που θα έχουμε. Ευχαριστούμε. Ο εισηγητής τώρα. Ένα-δύο λεπτά παρακαλώ. Α, μάλλον προηγουμένως, πριν ε, ο συντάκτης της νομοδότης πάρει το λόγο, εκπρόσωπος της ε, Ετέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ένα-δύο λεπτά δεν είναι πολύ για να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ε, όχι, δεν χρειάζεται να απαντήσετε στις ερωτήσεις, απλά να μας ε, παρουσιάσετε τη δήλωσή σας. Πολύ σύντομα, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον ε, σας στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Άικουτ και τους ε, σκιώδεις που παρουσίασαν τις απόψεις τους. θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι παρακολουθούμε την οικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνομιλούμε και με επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που φαίνεται και στην έκθεση επενδύσεών μας, την οποία σας συστήνω. Βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας και είναι πολύ ενδιαφέρουσα όσον αφορά τις προβλέψεις για την οικονομία. Θα ήθελα να πω ότι τέσσερι ε, τομεί προτεραιότητα έχουμε για να στηρίξουμε την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση σε κλιματική δράση, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσει, σε υποδομέ. Ε, και θα ήθελα να πω ότι στηρίζουμε την γεωγραφική ισορροπία, στηρίζουμε προγράμματα ανάπτυξης δυναμικού, παρέχουμε συμβουλές Όλα αυτά αποτελούν τμήμα του ε, επιχειρηματικού μοντέλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και ε, αυτό πολύ συχνά είναι σημαντική διαφορά για να μπορέσουν να απογειωθούν εντό εισαγωγικών τα προγράμματα. Ε, η μετατροπή σε κλιματική τράπεζα είναι πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική, αλλά νομίζω ότι είναι και λογική στους καιρούς που ζούμε. Πιστεύουμε επίσης ότι θα είμαστε ουσιαστικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην υποστήριξη της Πράσινης συμφωνία του Green Deal. Ήδη συνεργαζόμαστε πολύ καλά με την Επιτροπή Φοντερ Λάιεν όσον αφορά την ε, δίκαιη μετάβαση και νομίζω ότι θα τα δείτε όλα αυτά τους επόμενους, τις επόμενες εβδομάδες. Θα ήθελα να κλείσω επισημένοντας ότι το σχέδιο Juncker, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ε, είχε πολύ σημαντικό αντίκτυπο και με τρίσιμο αντίκτυπο Έχουμε ε, ένα πολύπλοκο σύστημα υπολογισμού του αντικτύπου. Το 2019, για παράδειγμα, δημιουργήσαμε πάνω από ένα εκατομμύριο θέσει απασχόληση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την διαφάνεια και τη σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρία πράγματα πολύ σύντομα. Πρώτον, ε, έχουμε πολύ σημαντική παρουσία στο Κοινοβούλιο. Πάντα είμαστε στη διάθεσή σας ε, για να έρθουμε να συνομιλήσουμε μαζί σας επίσης ευθυγραμμιζόμαστε απολύτως με τα πρότυπα που ανέφερε η κυρία Ομπρή. Και εγώ και οι συναδελφοί μου μπορούμε να ε, συναντηθούμε μαζί σα Είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφάνεια, τις μη συνεργάσιμε δικαιοδοσίε. Ε, δεν χρειάζεται να μας πείτε να τα κάνουμε αυτά, τα κάνουμε ήδη. Και η τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να στηρίξουμε και τις δικές εργασίες. Αν έχετε περισσότερε ερωτήσεις, σας παρακαλώ να με ενημερώσετε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ένα λεπτό έχετε, αν θέλετε τότε απλά να ευχαριστήσω ε, όλους τους ομιλητές και τους Ε, Νομίζω ότι στα περισσότερα θέματα μπορούμε να βρούμε μια λύση και όσον αφορά την ψηφιοποίηση και φυσικά διαβάσαμε την έκθεση επενδύσεων αλλά μετά από την ε, ε, προθεσμία κατάρτισης της γνωμοδότησης. Σίγουρα πάντως διαβάζουμε τις εκθέσεις σας όσον αφορά τα τις κοινωνικές πτυχές που αναφέρθηκαν. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να το συζητήσουμε και να βρούμε συμβασμό όσον αφορά την κλιματική τράπεζα. Να πω στο ECR ότι μιλάμε για δημόσια τράπεζα, δεν πρόκειται για ιδιωτική τράπεζα. Νομίζω ότι λογικά είναι πιο πολιτικοποιημένη, διότι αλλιώς γιατί να έχει κανείς μια δημόσια τράπεζα με δημόσιο χρήμα που είσαι σε αυτήν. Ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η ίδια θέλει να γίνει κλιματική τράπεζα. Βέβαια, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι καλή ιδέα αυτό, αλλά νομίζω ότι όλοι νιώθουν ότι είναι καλή ιδέα. Το, το, το πώ θα γίνει ακριβώ αυτό, η κοινωνική διάσταση, το Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση ε, είναι θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Άκουσα και αυτό που λέτε ότι είναι ήδη τέλεια τα θέματα όσον αφορά τη διαφάνεια, αλλά μπορεί να σας σπρώξουμε λίγο παραπάνω. Είχαμε και στο παρελθόν τη συζήτηση αυτή. Ε, σίγουρα όμως μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πάντω ε, προσβλέπω να λάβω τι ε, συμβαστικέ προτάσει ε, και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε ευρεία συνένεση πάνω στη γνωμοδότηση αυτή. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, μου φαίνεται και μένα ότι μπορούμε να έχουμε μια έκθεση που θα αφήσει ικανοποιημένου του περισσότερου. χρονοδιάγραμμα λοιπόν. 2 Δεκεμβρίου παρουσίαση τη νομοδότηση. Σε προθεσμία υποβολή τροπολογιών 9 Δεκεμβρίου. Εξέταση των ε, τροπολογιών 22-23 Ιανουαρίου. 6 Φεβρουαρίου ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ και ε, Ολομέλεια του Μαρτίου. Και 13 ε, Ιανουαρίου στο Στρασβούργο έχουμε σχετική ακρόαση. Ευχαριστώ τον εισηγητή και όλους τους κοιόδες εισηγητές ε, και περνάμε τώρα στα θέματα 6, 7 και 8. Πρόκειται για απαλλαγέ. Όποιος θέλει να αποχωρήσει, παρακαλώ να το κάνει αυτό ήσυχα. Ο uh, our μας είναι ο κύριος Epping αλλά τον αντικαθιστά ποιος ο κύριος Σιουτζικά οπότε παρακαλώ πέντε λεπτά αν τα χρειάζεστε Αλλιώ μην τα χρησιμοποιήσετε όλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όντω μιλάω εκ μέρου του κύριου Έπινγκ, ο οποίο ζητά συγγνώμη που αποσιάζει, αλλά δεν μπορούσε να έρθει σήμερα γιατί είχε ανελημμένε υποχρεώσει και μου ζήτησε να σα πω τα εξή. Θέλει πρώτα απ' όλα να σα ενημερώσει για τρία θέματα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη σήμερα για απαλλαγέ. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και πρόκειται και για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών όσον αφορά τους λογαριασμούς του 2018. Πρώτα απ' όλο ο κύριος Σέπινγκ θέλει να γνωστοποιήσει ότι κατά τη γνώμη του Λεκτικού Συνεδρίου οι πράξει τη ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, τη Αρχή Ασφαλή Παγκοσμίου Συντάξεων και τη Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών είναι κάθε, από κάθε ουσιώδη πλευρά νόμες και κανονικές. Για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών είχε κάποιε παρατηρήσει γιατί υπάρχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά ε, κάποιους ε, πόρους. Μιλώντας όμως με εκπροσώπους από ε, την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή των Αξιών και Αγορών φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ μικρές και ότι ο έλεγχος έγινε στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και εγκρίθηκαν και από την Ευρωπαϊκή Πετροπή και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Όλα καλά. Πάντως υπενθυμίζει ο κύριος Επίνγκ ότι έχουμε κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή ε, Τραπεζών διότι όλο και περισσότερο μεταφέρει το έργο της και τα καθήκοντά της ε, από τις ε, ε, από τις, τα καθήκοντά της τα αρχικά προς άλλα καθήκοντα και πρέπει να σεβαστούμε την ανεξαρτησία. Ο κύριος Έπινγκ θέλει να πει ότι μπορούν να υπάρξουν οικονομίες κλίμακας που δεν έγιναν όμως λόγω ανεπαρκούς χρήσης των κοινών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων της ε, αρχής ε, τραπεζών και της αρχής ε, κινητών αξιών και αγορών. Και έτσι καλεί την Αρχή Τραπεζών ενισχύσει την συνεργασία τη με την ΕΑΚΑ στον τομέα των υπηρεσιών διοικητική υποστήριξη και των υπηρεσιών διαχείριση εγκαταστάσεων, οι οποίε βέβαια δεν σχετίζονται με τι βασικέ δραστηριότητε. Όσον αφορά την ΕΙΟΠΑ, ο κύριο Επίνγκ θέλει να υπογραμμίσει ότι όλες οι αρμοδιότητες προχωρούν και τηρούνται εντός προθεσμίες και ότι θα πρέπει να φροντίσει η ΟΠΑ να παραμείνει στην εντολή που της έχει ανατεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπως ισχύει και για τις άλλες αρχές, έτσι και για την αρχή ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων, ε, περνάει από την ρύθμιση στην εποπτεία. Το 2018 λοιπόν ε, είναι η απαλλαγή από εμά για τις τρεις αυτές αρχές όσον αφορά του λογαριασμού του 2018, αλλά να κοιτάξουν οι αρχές το ρυθμιστικό του έργο. Ο κύριο Έμπικ επίσης προσβλέπει σε επικοδομητική συνεργασία με τους Κιώδης και σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Όντως αντικαταστήσατε πάρα πολύ καλά τον κύριο Έπινγκ θα έπρεπε να είχα πει ότι η συγκητή είναι ο κύριος Σινιέσκη γιατί πρόκειται για γνωμοδότησή μας στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Ο κύριος Φερνάντες έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι εδώ ο σκιώδης συγκητής μας, αλλά μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω εγώ. Και θα σας διαβάσω τι μου έδωσε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή μας για το έργο του για τους τρεις φακέλους. Εξε, εκ μέρους της ομάδας των σοσιαλδημοκρατών θέλουμε να πούμε ότι στηρίζουμε τις ιδέες του παρόλο που έχουμε και άλλες ιδέες για να ενισχύσουμε περισσότερο το κείμενο. Πρώτον, θέλω να μιλήσω για τον κεντρικό ρόλο των αρχών υπέρ του, της σταθερότητας του οικονομικού μας συστήματος και πέντε διαφάνειες. Δεύτερον, θέλω να υποβάλω κάποιες τροπολογίες για να τονίσω τη σημασία που έχει η εποπτεία του δημόσιου οικονομικού τομέα και την καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων παράνομες δραστηριότητες αλλά και τη διαφθορά. Είναι πολύ βασικό η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να φροντίζει για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητε ή από την τρομοκρατία. Για τις άλλες δύο αρχές, την ΕΣΠΑ και την ΙΟΠΑ, πρέπει να συνεχίσουν αποτελεσματικά να τελούν το έργο τους. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει μια ανοιχτή και ανεξάρτητη δίκηση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να επικεντρωθούμε στα συμφέροντά μας υπέρ ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας. Ευχαριστώ πολύ που σημειώσατε τις προτάσεις αυτές. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για το Renew. Ζωέμποε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για τη δουλειά του την χάνει να είμαι σκιώδης εισηγητής στην Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών για την απαλλαγή της ΕΙΟΠΑ και της ΕΒΑ. Αλλά εδώ θα μιλήσω από την ιδιότητα του μέλους της ε, Επιτροπής ΕΚΟΝ λαμβάνοντα υπόψη όλε τι νομικέ ε, πτυχέ του θέματο έχω σκοπό να υποβάλω τρει τοπολογίε στι τρει εκθέσει για να εκφράσω κάποιε διαφορετικέ απόψει. Σε σχέση με αυτό που ονομάζεται δίκαιη επιστροφή των ε, δημοσιονομικών συνεισφορών των κρατομελών, δεν μου φαίνεται αυτό συμβατό με την οικοδόμηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον όπω την αντιλαμβανόμαστε, ή όπω εμεί την αντιλαμβανόμαστε τέλο πάντων, και διερωτώ και για του πόρου που αποδίδονται στου τρει οργανισμού σε σχέση με τι αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί. Απαντώντα και στα ερωτήματα που τους έχουν τεθεί για την εκτέλεση ε, των εργασιών τους. Ε, για τις μετακυλήσεις συνεχώς ε, τίθενται ερωτήματα, υπάρχουν αναβολές και καθυστερήσει, οπότε Είμαι υπέρ τη ε, καλή διαχείριση των πόρων, αλλά πραγματικά διαρωτώ με μήπω κάποιε φορέ ε, ζητάμε το ανέφικτο από αυτού του οργανισμού. Δηλαδή να κάνουν περισσότερα χωρί να αυξηθούν οι πόροι και όσα διαθέτουν. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν αυτό ισχύει, κατά πόσο η πολιτική μα είναι ε, βιώσιμη και θα του επιτρέψει να λειτουργούν και στο μέλλον. Και ω συνέπεια τη πρώτη ερώτηση για τη χρήση των ε, την πρόσληψη των συμβασιούχων υπαλλήλων. Ε, δεν έχω καμία αμφιβολία για την ποιότητα τη εργασία του, όμω ε, είναι μια λύση που ίσω να μην είναι καλύτερη, ακόμη και αν ε, βραχυπρόθεσμα είναι η λιγότερο δαπανηρή. Πρέπει να κοιτάξουμε και το μέλλον και στον τομέα της πληροφορικής ας πούμε έχουμε μία ε, εξάρτηση, σχέση εξάρτησης διαρκείας κι όμω, ο τομέα τη πληροφορική είναι ζωτική σημασία την επιβίωση των οργανισμών και θα πρέπει να επενδύσουμε ενδεχομένω μακρο... πιο μακροπρόθεσμα στο προσωπικό που προσλαμβάνουμε. Εάν θέλουμε να είμαστε συνεπεί απέναντι στου πολίτε που δικαίω μα ερωτούν για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των ευρωπαϊκών οργανισμών, εάν θέλουμε να επιδείξουμε συγκεκριμένα επιτέγματα, πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ, διότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί εποπτεία εκτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο. Τα όσο αναλαμβάνουν αυξανόνται κάθε χρόνο, όμω δεν παίρνουν και του πόρους. πόρου. Μόνο τέσσερις επιπλέον θέσεις προσφέρθηκαν για τις νέες ε, ευθύνες ε, τις νέες ευθύνες του ε, ΕΜΠΑ, της ΕΜΠΑ, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, κάτι που, κακώς είναι, που προφανώς είναι μήνυμα ως προς τις κοινωνικές προτεραιότητες, ιδίως ήταν η Deutsche Bank, η Δανέζικη τράπεζα προχώρησε σε έρευνες για τη λεύκανση. Εμπλέκονταν δύο τραπεζικά εντρέματα και δύο οργανισμοί ανεξάρτητοι, εξωτερική υπεργολαβία. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκίγκολτ, την ο συγκεκριτής των Πρασίνων. So, thank you Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ερήμην του και τον κύριο Έπινγκ που ήταν ο θεματοφύλακας ε, της δουλειάς της γραμματείας και επίσης που τόνισε τα θέματα που έθιξε και το ελεγκτικό συνέδριο. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την γραμματεία και τους συνεργάτες που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Ε, να ακολουθεί κανείς ε, πιστά την εντολή του ε, είναι για μένα αστικός μύθος ε, του Παρισιού, του Λονδίνου και της Φραγκφούρτης, διότι κανείς δεν μπορεί ακόμα να αποδείξει ότι ξεπέρασαν τα όρια της εντολής τους. Αντιθέτως, έχουμε πολλούς τομείς και ο κ. Μπουγιά αναφέρθηκε σε κάποιους από αυτούς, όπου δεν είχαν αρκετούς πόρους να κάνουν αυτά που τους αναθέσαμε. Εγώ ψάχνω Λοιπόν, ακόμη παράδειγμα ε, όπου οι ESA ε, να έχουν ξεπεράσει τα όρια της θητείας τους. Για μένα είναι σαν τους κροκοδίλους στους υπονόμους της Νέας Υόρκης. Και εγώ δεν καταλαβαίνω το θέμα των πλεονασμάτων. Ε, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, το πρόβλημα λύθηκε το 2012. Το πώς ε, ξαναπροέκυψε δεν ε, το καταλαβαίνω, θα ήθελα πολύ να το καταλάβω. Επίσης, όσον αφορά τις ρυθμίσεις μικτής ε, χρηματοδότησης, συμφωνώ ότι αποτελούν πρόβλημα για την ανεξαρτησία, την αυτονομία των αρχών εποπτείας, διότι κάποιοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να είναι αυτόνομος φορέας, εγώ όμως διαφωνώ, διότι η μελλοντική πρόοδος τους εξαρτάται από ε, επιπλέον χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι ο λόγος που έχουμε τόσα προβλήματα όσον αφορά την ε, απόκτηση επαρκών πόρων. Πάντως, ε, ή θα πρέπει να έχουμε μια αμφίσιμη διάταξη ή θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να την ε, διαγράψουμε. Συμφωνώ και με τον κύριο Ποχέ όσον αφορά το ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τις ε, αρχές εποπτείας ε, να κάνουν περισσότερα ε, όσον αφορά την νομοποίηση παράνομων εσόδων. Ε, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, φαίνεται όμω ότι τώρα έχουν επαρκή χρηματοδότηση. Είχαμε πρόσφατα και το σκάνδαλο της Danske Bank, το οποίο θα πρέπει να θεωρηθεί σαφής αποτυχία ε, διακυβέρνησης και μάλιστα όχι από το 2014, ωστόσο δείχνει ότι υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν προβλήματα στη διακυβέρνηση και η ε, πολύτιμη δουλειά που έκανε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ε, ε, πέρασε στο ράφι χωρίς επαρκή εξέταση και έτσι και έτσι έχασε μέρος του γοήτρου του της και το σώμα των επόπτων Ε, το ότι το επέτρεψε το σώμα των επόπτων χωρί αρκετού ε, αυστηρούς κανόνες, αυτό δεν είναι αρκεί για μας. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν προκύψει με τις ε, αρχές εποπτείας. Πάντως προσβλέπω στη συνέχεια των εργασιών. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ Σβέν. Εγώ είμαι ο μόνος που μπορώ να πάρω το λόγο στη διαδικασία Catch the Eye, αλλά δεν πειράζει. Δεν, θα μπορώ να παραιτηθώ από το δικαίωμα αυτό. Δεν ξέρω αν ε, θέλει να συμπληρώσει κάτι ο εισηγητή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις σημαντικές παρατηρήσεις τους ε, και ε, υπόσχομαι να τις μεταφέρω στον κύριο Έπινγκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να συνοψίσω το χρονοδιάγραμμα. Εξέταση των τροπολογιών 22-23 Ιανουαρίου. Ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ την ίδια μέρα. Ψηφοφορία στην ΚΟΝΤ 19-20 Φεβρουαρίου. Δεύτερη ολομέλεια του Μαρτίου. Αυτά για σήμερα. Ε, νομίζω ότι είχαμε ενδιαφέρον ε, απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Καλό σας βράδυ.